Okay, good morning everybody. Καλημέρα σας. Θα μιλήσω σουηδικά. Επομένως, φορέστε σας παρακαλώ πολύ τα ακουστικά σας. Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω σε αυτή την τελευταία συνεδρία της Επιτροπής μας πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Σημείο 1 της ημερήσιας διάταξης, έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Θα ήθελα να σας ενημερώσω για το ότι το σημείο 8 της ημερήσιας διάταξης, ψηφοφορία για την γνωμοδότηση της κυρίας Κράτσα, το σημείο αυτό θα αναβληθεί για τις 3 Σεπτεμβρίου. Ελπίζω να μην υπάρχει κάποια αντίρρηση στην αλλαγή αυτή και αν δεν υπάρχει κάποια αντίρρηση τότε μπορούμε να εγκρίνουμε την τροποποιημένη ημερήσια διάταξη. Περνάμε λοιπόν στο σημείο 2 της ημερήσιας διάταξης. Ανακοινώσεις του Προέδρου σχετικά με τις συστάσεις των συντονιστών. Λάβατε τα πρακτικά από τη συνεδρίαση των συντονιστών. Δεν έχουν επέλθει κάποιες αλλαγές, ούτε έχουν προταθεί κάποιες αλλαγές, επομένως μπορούμε να εγκρίνουμε και τα πρακτικά αυτά. Περνάμε στο σημείο 3 της ημερήσιας διάταξης. Ανακοινώσεις του Προέδρου. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι αύριο αύριο στις 9 το πρωί η Λέιλα Ζανά Κούρδη από την Τουρκία θα είναι μαζί μας και θα έχουμε μια κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όπως γνωρίζετε πρόκειται για μια πρωτοβουλία της δικής μας Επιτροπής και πραγματικά ελπίζω ότι θα έρθουν στη συνεδρίασή μας όσο δυνατόν περισσότεροι ευρωβουλευτές αύριο το πρωί όταν η Λίλα Ζανά έρθει να μας μιλήσει για την ελευθερία της έκφρασης και τα δικαιώματα των γυναικών στην Τουρκία. Ας συνεχίσουμε λοιπόν τώρα με τη μερίσια διάταξη. Περνάμε στο βασικό σημείο της σημερινής ημερήσιας διάταξης, σημείο 4 στο σημείο αυτό. Θα ήθελα να καλωσορίσω πολύ θερμά τους εκπροσώπους της Κυπριακής Προεδρίας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε τις απόψεις σας. Είχα τη δυνατότητα να σας συναντήσω όταν πήγαμε ως αντιπροσωπεία στην Κύπρο. Είναι ένα καταπληκτικό πανέμορφο νησί. Είχαμε πολύ ωραίες συναντήσεις και πολύ ωραίες συνεδριάσεις και θα ήθελα πραγματικά να ακούσω τι σχεδιάστε στα πλαίσια της Κυπριακής Προεδρίας. Ξέρω ότι ενδιαφέρεστε πάρα πολύ για τα ζητήματα της ισότητας, πάρα πολύ σημαντικά για τη δική μας την Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Θα ασχοληθούμε με ζητήματα όπως τα δικαιώματα των γυναικών προφανώς, αλλά και την βία κατά των γυναικών που διαπράτεται από άντρε. Και αυτό είναι το ζήτημα το οποίο μας απασχολεί και πιστεύω ότι θα πρέπει να μας απασχολήσει και τους επόμενους έξι μήνες και θα έχουμε μια πολύ επικοδομητική συνεργασία προκειμένου να καταφέρουμε να σημειώσουμε σημαντική πρόοδο στα ζητήματα αυτά στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταρχάς θα ήθελα να δώσω το λόγο στους υπουργούς. Ο καθένας σας διαθέτεται από 20 λεπτά, με 20 λεπτά και οι δύο μαζί, με συγχωρείτε λέει ο πρόεδρος, 20 λεπτά και οι δύο μαζί. Θα δείτε λοιπόν πώς θα διαχωρίσετε το χρόνο αυτό και αφού ολοκληρώσετε τις παρεμβάσεις σας, θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε τους συντονιστές της Επιτροπής μας και στη συνέχεια ενδεχομένω να πάρουν το λόγο και άλλα μέλη τη Επιτροπή μα. Και στη συνέχεια θα έχετε προφανώ τη δυνατότητα να απαντήσετε σε ενδεχόμενε ερωτήσει. Για άλλη μια φορά θα ήθελα να σας καλωσορίσω πολύ θερμά στην Επιτροπή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ και σας δίνω ευθύ αμέσως το λόγο. Αποφασίστε εσείς που θα ξεκινήσει πρώτος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αποτελεί για μένα τιμή που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας η Κυπριακή Προεδρία αναγνωρίζει τον ενισχυμένο ρόλο του Κοινοβουλίου, το οποίο θεωρεί σύμμαχό της στις προσπάθειες για πρόοδο και ανάπτυξη στην Ευρώπη. Η ισότητα ανδρών και γυναικών αποτελεί θεμελιώδη αρχή και κοινή αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενσωματωμένη στην Ευρωπαϊκή Συνθήκη Εγκαθίδρυσης. Η Κύπρος παραμένει δεσμευμένη στην αρχή της ισότητας και είναι έτοιμη να συμβάλλει με όλες τις δυνάμεις στην προώθηση της εφαρμογής της διακήρυξης για τα δικαιώματα των γυναικών, της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Ισότητα και του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών. Παράλληλα, όπως όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κύπρος είναι προσιλωμένη στην εφαρμογή του προγράμματος δράσης και διακήρυξης του Πεγίνου, το οποίο εξακολουθεί να αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό καθοδηγητικό εργαλείο για την προώθηση της ισότητας στις κοινωνίες μας. Επίσης, στα πλαίσια της στρατηγικής Ευρώπη 2020, η ισότητα ανδρών και γυναικών αναδεικνύεται ως απαραίτητη προϋπόθεση για την προώθηση της εφαρμογής της, καθότι σχετίζεται άμεσα με τους στόχους της απασχόλησης, της ισομισθίας, της συμφιλίωσης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, της αναβάθμισης των υπηρεσιών φροντίδας παιδιών και άλλα. Όλα τα προαναφερθέντα συνηγορούν στο ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου διαπερνά οριζοντίως όλους τις τομείς, τους τομείς της ζωής και η επίτευξή της προϋποθέτει τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων περιλαμβανομένων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Ω γνωστό, τον Οκτώβριο του 2011 η Κύπρος με τη Δανία και την Πολωνία υιοθέτησαν μία κοινή διακήρυξη η οποία εκφράζει τις προτεραιότητες και τις δεσμεύσεις των τριών χωρών για την επίδευξη της ισότητας των φύλων κατά τη διάρκεια της 18μηνης Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη σημερινή παρουσίαση ενώπιον της Επιτροπής σας θα επικεντρωθώ στο θέμα της βίας κατά των γυναικών, της ισόρροπης συμμετοχής ανδρών και γυναικών στις θέσεις λήψεων αποφάσεων και πιο συγκεκριμένα στα διοικητικά συμβούλια των εταιριών, στο, θέμα γυναίκες και οικονομική κρίση, στο νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020 και στην χρηματοδότηση προγραμμάτων για θέματα ισότητας και βίας κατά των γυναικών καθώς και στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ισότητας των Φύλων. Θα ξεκινήσω με τη βία κατά των γυναικών. Αξιοπρέπεια, ακαιρεότητα και τέλος τη βία λόγω φύλου είναι ένας από τους πέντε τομείς προτεραιότητας που καθορίζονται στη στρατηγική που εκπώνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς και στη διακήρυξη για τα δικαιώματα των γυναικών. Το Συμβούλιο, το οποίο θεωρεί το θέμα αυτό ως προτεραιότητα, ζήτησε τη λήψη κατάλληλων μέτρων, τα οποία μάλιστα περιλαμβάνονται στο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων 2011-2020. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει ενεργά μέτρα για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και έχει μάλιστα καλέσει την Επιτροπή να αναπτύξει στρατηγική για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και να καθιερώσει ένα ευρωπαϊκό έτος αφιερωμένο στο πρόβλημα αυτό. Στον τομέα αυτό το Συμβούλιο συνεργάζεται στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για σχετικές προτάσεις συμπεριλαμβανομένης της πρότασης κανονισμού για την αμοιβαία αναγνώριση των μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις, η οποία συμπληρώνει την οδηγία για το Ευρωπαϊκό Διάταγμα Προστασίας. Η πρόταση αυτή είναι πολύ σημαντική για τους Ευρωπαίους πολίτες, εφόσον θα ολοκληρώσει το νομικό πλαίσιο προστασίας των θυμάτων παρέχοντας ένα γρήγορο και εύκολο μηχανισμό διασυνοριακής αναγνώρισης των μέτρων για την προστασία των ατόμων αυτών η Κυπριακή Προεδρία, αναγνωρίζοντα τη σημασία που έχει η πρόταση αυτή για τα θύματα, στοχεύει στην ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων στο Συμβούλιο. Παράλληλα, στα πλαίσια εφαρμογή του προγράμματο δράση του Πεκίνου, η Κυπριακή Προεδρία εργάζεται πάνω στο προσχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου με θέμα καταπολέμηση τη βία κατά των γυναικών, υπηρεσίε υποστήριξη θυμάτων ενδοοικογενειακή βία, το οποίο βασίζεται στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Ισότητας των Φύλων. Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφωνούν για την ανάγκη καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών. Στο παρελθόν έχουμε ήδη συνεργαστεί με επιτυχία για την δημιουργία και προώθηση του προγράμματος Δάφνη, της Οδηγίας για την Εμπορία Προσώπων και της Οδηγίας για το Ευρωπαϊκό Διάταγμα Προστασίας. Είναι με ευχαρίστηση που αναφέρω ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση με το Ευρωκοινοβούλιο όσον αφορά την οδηγία για την προστασία των θυμάτων, στην οποία μάλιστα ενσωματώνεται και η διάσταση του φύλου. Η Κυπριακή Προεδρία θα επικεντρωθεί στο θέμα των υπηρεσιών στήριξη θυμάτων ενδοικογενειακή βία, αναπτύσσοντα μάλιστα δείχτε στα πλαίσια προγράμματο δράση του Πεκίνου. Όπως και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο ζήτησε την δημιουργία ευρωπαϊκής στρατηγικής για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Αλλά εναπόκειται στην Επιτροπή να αποφασίσει αν και πότε θα προχωρήσει στο σχεδιασμό, στο σχεδιασμό μιας τέτοιας στρατηγικής. Η Κυπριακή Προεδρία θα προωθήσει την ανάπτυξη μακροπρόθεσμης επιχορηγημένης και συντονισμένης ευρωπαϊκής διαφωτιστικής εκστρατείας για τη βία κατά των γυναικών στοχεύοντας διάφορες ομάδες περιλαμβανομένων ανδρών και αγοριών και εμπλεκόμενες γυναικείες οργανώσεις και εμπλέκοντας γυναικείες οργανώσεις και άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις. Θα προωθηθεί επίσης η καθιέρωση του 2015 ως Ευρωπαϊκού Έτους Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών. Ισόρροπη συμμετοχή ανδρών και γυναικών στις θέσεις λήψεως αποφάσεων στα διοικητικά συμβούλια των εταιριών. Οι γυναίκε ενώ αντιπροσωπεύουν πέρα του 60% των νέων απόφοιτων πανεπιστημίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υποεκπροσωπούνται σημαντικά στις θέσεις λήψης αποφάσεων στην δημόσια και οικονομική ζωή. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Ιανουάριο του 2012, μόνο το 14% περίπου των μελών των διοικητικών συμβούλων και μόλις το 3% των προέδρων διοικητικών συμβουλίων των μεγάλων εταιριών, εισηγμένο στα χρηματιστήρια των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν γυναίκες. Η Επιτροπή, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, δήλωσε ότι θα αντιμετωπίσει την ανισορροπία αυτή μέσω στοχοθετημένων πρωτοβουλειών. Μάλιστα, η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, κυρία Ρέντινγκ, με δική της πρωτοβουλία ζήτησε από τις εταιρείε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να υπογράψουν μια δέσμευση σύμφωνα με την οποία μέχρι τον Μάρτιο του 2012 δεσμεύονται θελοντικά να αυξήσουν την παρουσία των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια τους μέχρι το και 30% έως το 2015 και 40% μέχρι το 2020. Στις 17 Φεβρουαρίου 2012 το Συμβούλιο Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, υγεία και Καταναλωτών διεξήγαγε συζήτηση με θέμα γυναίκε στα διοικητικά συμβούλια των εταιρεών μελετώντα τρόπου βελτίωση του προβλήματο. Ορισμένοι υπουργοί υποστήριξαν τη χρήση δεσμευτικών ποσοστώσεων, ενώ άλλοι, πολλοί άλλοι, τάχθηκαν υπέρ τη εθελοντική προσέγγιση, τουλάχιστον στο παρό στάδιο. Μετά τη συζήτηση, η Επιτροπή δρομολόγησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με πιθανά μέτρα, η οποία έκλεισε στις 28 Μαΐου. Η Επιτροπή εξετάζει τώρα κατά πόσον θα προτείνει νομοθετική πρωτοβουλία για την διασφάλιση της ισόρροπης συμμετοχής ανδρών και γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των εταιριών. Τα βασικά μηνύματα είναι ότι το Συμβούλιο υποστηρίζει τη γενική ιδέα της ισότιμης συμμετοχής ανδρών και γυναικών στις θέσεις λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα και όλους τους τομείς, προκειμένου να γίνεται αξιοποίηση όλων των ταλέντων και των δεξιοτήτων ανδρών και γυναικών. Αναγνωρίζεται συνεχώς ότι η ισότητα ανδρών και γυναικών επιφέρει οικονομικά ωφέλη μέσω της αύξησης της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και επίσης οδηγεί σε καλύτερες αποφάσεις για πιο στενές και δυνατές, πιο δυνατές επιχειρήσεις. Το να μην δίδεται η ευκαιρία στι γυναίκε να χρησιμοποιούν τα ταλέντα του είναι άδικο και συνιστά σπατάλη ανθρώπινου κεφαλαίου, κάτι που η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να χάνει. Οι Υπουργοί συζήτησαν το θέμα της, ισορροπία της ισορροπίας μεταξύ των φύλων στα διοικητικά συμβούλια των εταιριών στο Συμβούλιο του Φεβρουαρίου. Υπάρχει ευρία αναγνώριση της ανάγκης να βελτιωθεί το ισοζύγιο της συμμετοχής ανδρών και γυναικών στη λήψη ε, επιχειρηματικών αποφάσεων. Ωστόσο, διάφορες χώρες έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Όπως γνωρίζετε, το Συμβούλιο δύναται να ενεργεί υπό την νομοθετική του ιδιότητα μόνο εφόσον υποβληθεί σχετική πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είμαστε σε αναμονή. Γυναίκες και οικονομική κρίση. Το 2009 στο πλαίσιο ετοιμασία τη στρατηγική Ευρώπη 2020, το Συμβούλιο υιοθέτησε μια σειρά συμπερασμάτων με θέμα την ισότητα των φύλων, ενδυναμώνοντα την ανάπτυξη και την απασχόληση, συμβολή στην μετά το 2010 στρατηγική της Λισαβόνας. Στα συμπεράσματα τονίζεται ότι η ισότητα των φύλων είναι ζωτική σημασία για την εκπλήρωση των στόχων τη Ευρωπαϊκή Ένωση για οικονομική και κοινωνική συνοχή, την επίτευξη ενός ψηλού επίπεδου απασχόλησης, τη διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας, αλλά και για την αντιμετώπιση των ευρύτερων δημογραφικών προκλήσεων. Ισχύουσα κατάσταση, η σημασία της ισότητας των φύλων με ευρύτερο οικονομικό πλαίσιο αναγνωρίζεται στη Στρατηγική Ευρώπη 2020 η οποία θέτει ως έναν από τους βασικούς στόχους την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης ανδρών και γυναικών ηλικίας 20 μέχρι 64 σε 75%. Σύμφωνα με το έγγραφο εργασία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τίτλο «Προόδος στον τομέα τη ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών το 2011, το 2010 το ποσοστό απασχόληση των ανδρών ήταν 75% ενώ το ποσοστό απασχόλησης για τις γυναίκες ήταν μόλις 62,1%. Η αύξηση του ποσοστού απασχόλησης των γυναικών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπης 2020. Η προώθηση της ισότητας δεν μπορεί να εκλαμβάνεται ως οικονομική επιβάρηση αλλά ως προϋπόθεση ζωτικής σημασίας για μια ισχυρή οικονομία όπου όλοι οι πολίτες μπορούν να συνεισφέρουν. Το Συμβούλιο αναγνωρίζει τη σημασία της ισότητας ανδρών και γυναικών στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης και την ανάγκη ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στη στρατηγική Ευρώπη 2020. Το Συμβούλιο υποστηρίζει τους στόχους της Βαρκελόνης για διευκολύνσεις στην παροχή υπηρεσιών φροντίδας παιδιών καθώς και άλλα σχετικά μέτρα όπως την καταπολέμηση των στερεοτύπων, τη σμίκριση του χάσματος αμοιβών μεταξύ αντρών και γυναικών, την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, στην επιχειρηματικότητα και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Το ζήτημα γυναίκα και οικονομική κρίση πρέπει να εξετάζεται σφαιρικά, προάγοντας την ισότητα είναι επίσης ένας τρόπος για την επίτευξη της δημοσιονομικής ισορροπίας την καταπολέμηση της φτώχειας, την αξιοποίηση των ταλέντων και δεξιοτήτων των γυναικών, ιδιαίτερα μέσα στα πλαίσια της πράσινης οικονομίας. Η ισότητα αποτελεί ένα ιδιαίτερο σημαντικό κεφάλαιο μέσα στο πλαίσιο των ευρύτερων δημογραφικών προκλήσεων. Όσον αφορά το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020, το πρόγραμμα Δάφνη που καταρτίστηκε από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με στόχο μεταξύ άλλων την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών τερματίζεται περί τα τέλη του 2013. Ένα διάδοχο πρόγραμμα έχει προταθεί από την Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια 2014-2020 το οποίο θα ενσωματώσει το μέρος και την ισότητα των φύλων του προγράμματος για την απασχόληση και την κοινωνική αλληλεγγύη. Το Συμβούλιο κατέληξε στις 8 Ιουνίου 2012 σε μερική γενική προσέγγιση επί της σχετικής πρότασης κανονισμού. Στο κείμενο περιλαμβάνεται σαφώς και η χρηματοδότηση δράσεων που να καλύπτουν και θέματα της διάστασης των δύο φύλων αλλά και της προστασίας των θυμάτων. Το Συμβούλιο και οι χώρες μέλη του Τρίου έχουν εκφράσει ξεκάθαρα τη δέσμευσή τους για την ισότητα των φύλων και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Όπως υπογράμμισε το Κοινοβούλιο στο πρόσφατο ψήφισμά του για το πρόγραμμα Δάφνη, είναι σημαντικό να συνεχιστεί η διαφώτιση και η ευαισθητοποίηση στον τομέα αυτό. Τρέχουσες προκλήσεις περιλαμβάνουν τον ακροτηριασμών των γυναικείων γεννητικών οργάνων, τα λεγόμενα εγκλήματα τιμή και του κινδύνου που αντιμετωπίζουν οι έφηβοι και τα παιδιά. Το Συμβούλιο και το Ευρωκοινοβούλιο έχουν κοινή ευθύνη να διασφαλίσουν ότι η ισότητα των φύλων παραμένει προτεραιότητα παρά τι περικοπέ των προπολογισμών. Η Κυπριακή Προεδρία θα συνεχίσει να προωθεί τη διασφάλιση τη διάσταση του φύλου και την καταπολέμηση τη βία κατά των γυναικών, δίνοντα ιδιαίτερη έμφαση στο σημαντικό ζήτημα των υπηρεσιών στήριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακή βίας. Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ισότητας των Φύλων. Η γενική στόχη του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Ισότητας των Φύλων είναι να συμβάλλει στην ενίσχυση και την προώθηση της ισότητας των φύλων, να ενισχύσει τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, στον αγώνα για για καταπολέμηση των διακρίσεων λόγου φύλου και να αυξάνει διαρκώς τη διαφώτιση γύρω από αυτά τα θέματα. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο έχει αναλάβει το ρόλο της υποστήριξης της, στις διαδοθικές προεδρίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά θέματα που άπτονται της παρακολούθησης του προγράμματος δράσης του Πεκίνου. Μέσα στα, πλαίσια, μέσα στα ευρύτερα πλαίσια των δημοσιονομικών περικοπών και της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης ο προπολογισμό του Ινστιτούτου έχει, έχει σημειώσει μείωση. Αναμένεται επίση ότι το Ινστιτούτο θα πρέπει να μειώσει το προσωπικό του κατά 5% τα επόμενα 5 χρόνια. Η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Ισότητα των Φύλων αποτελεί παράδειγμα τη κοινή δέσμευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προώθηση, για την προώθηση της των φύλων. Η ύπαρξη διαθέσιμων συγκρίσιμων στατιστικών στοιχείων κατά φύλου αποτελεί απαραίτητη προπόθεση για τη χάραξη ορθών πολιτικών ισότητα των φύλων, ενώ το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο έχει καταστεί σε σύντομο χρονικό διάστημα ένα κέντρο <clears throat> με μεγάλη εμπειρία στον τομέα αυτό. Η αξία του έργου του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου δεν θα πρέπει να τεθεί υπό αμφισβήτηση μέσα στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης. Η Κυπριακή Προεδρία είναι ευγνώμων για τη συνεργασία της με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ισότητας των Φύλων, το οποίο ετοίμασε έκθεση για τις υπηρεσίες στήριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, θέμα το οποίο έχει επιλεγεί για να αποτελέσει το αντικείμενο των συμπερασμάτων του Συμβουλίου που έχω ήδη αναφέρει. Όσον αφορά τις δράσεις τις οποίες έχει καθορίσει και προγραμματίσει η Κυπριακή Προεδρία, να σας αναφέρω ότι θα διοργανωθεί ε, θα, θα λάβει η χώρα διοργάνωση Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Υψηλού Επιπέδου με θέμα την ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών στα πλαίσια του οποίου θα παρουσιαστεί η πρόοδος που σημειώθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και άλλες πρακτικές που εφαρμόζονται στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες στον τομέα αυτό. Το συνέδριο αυτό θα γίνει στη Λευκοσία στις 8 και 9 Νοεμβρίου 2012 και ελπίζουμε να έχουμε και τον πρόεδρο της Επιτροπής ΦΑΜ για να ακούσουμε απευθείας τις απόψεις του. Επίσης θα γίνει θα φιλοξενηθεί η Επιτροπή Υψηλού Επιπέδου για την Ενσωμάτωση της Διάστασης του Φύλου στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, η οποία διασφαλίζει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα ισότητας ανδρών και γυναικών. Αυτά, αυτές οι δύο συναντήσεις θα γίνουν από το Υπουργείο Δικαιοσύνη της Κύπρου. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι θα ενημερώσει και η συνάδελφος για τη δική της συνάντηση που θα γίνει στην ε, Λευκοσία. Κυρίες και κύριοι, κλείνοντα θέλω να επαναλάβω τη σημασία που αποδίδει η Κυπριακή Προεδρία στη συνεργασία της με το Ευρωκοινοβούλιο και ευελπιστώ στην ενίσχυσή της στα πλαίσια της εξάμηνης Προεδρίας μας. Ευχαριστώ για την προσοχή σας και μετά την παρουσία της αγαπητής συναδέρφου θα είμαι στη διάθεσή σας για οποιασδήποτε διευκρινήσεις ή παρατηρήσεις. Ευχαριστώ. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, αποτελεί πραγματικά μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή για μένα στα πλαίσια της άσκησης της εξάμενης Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία να βρίσκουμε σήμερα μαζί με τον συνάδελφο Υπουργό Δικαιοσύνη και Δημόσια Τάξη για να καταθέσουμε τι σκέψει αλλά και τι προτεραιότητε τη Κυπριακή Προεδρία σε ένα κεφάλαιο το οποίο είναι καθοριστικό για την πορεία τη Ένωση μα. Και είναι με χαρά που ε, βρίσκομαι εδώ για να υπογραμμίσω την τεράστια σημασία που έχει η συνεργασία μαζί σας σε αυτό το μεγάλο κεφάλαιο. Κατά τη διάρκεια τη επίσκεψη τη επιτροπή ε, στην Κύπρο είχαμε τη δυνατότητα να σα ενημερώσουμε τόσο για το πρόγραμμα τη Κυπριακή Προεδρίας αλλά και για την κατάσταση στα ζητήματα της ισότητα στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ελπίζω ότι η επίσκεψη ήταν επωφελής, απολαύσατε την Κυπριακή φιλοξενία και είμαι σίγουρη ότι στα πλαίσια της άσκησης της εξάμενης Προεδρίας θα έχουμε ξανά τη χαρά να σας φιλοξενήσουμε στην Κύπρο. Από τη δική μου την πλευρά θέλω να πω ότι ήταν μια εξαιρετικά χρήσιμη και επικοδομητική συνάντηση. Επιτρέψτε μου να επισημάνω ότι η Κυπριακή Προεδρία στηρίζεται στη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να δουλέψουμε προς την κατεύθυνση της υλοποίησης των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο τη διασφάλιση ψηλού επίπεδου ποιότητας ζωής για κάθε πολίτη της Ένωσης. Ενδεικτικό της σημασίας που αποδίδουμε στο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι το γεγονός ότι αρχίσαμε από τον Νοέμβριο τις επαφές με ευρωβουλευτές, μέλη των αρμόδιων επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στο πλαίσιο αυτό είχα την ευκαιρία να συναντήσω τον Πρόεδρο, τον αγαπητό κύριο Γκούστασον, αλλά και τους συντονιστές των ομάδων των πολιτικών κομμάτων. Οι συναντήσεις αυτές ήταν ιδιαίτερα εποφιλείς, αφού είχαμε την ευκαιρία να ενημερωθούμε για τις θέσεις του Κοινοβουλίου σε πολλά από τα θέματα που θα κληθούμε να χειριστούμε ως Κυπριακή Προεδρία. Αναλαμβάνουμε την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για την Ευρώπη. Η κρίση έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των πολιτών. Είναι πολλές οι πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα πλήστα κράτη σε σχέση με την κοινωνική πολιτική και την πολιτική απασχόληση. Ένα από τα μεγαλύτερα διακυδεύματα σε περιόδους κρίσης είναι η πορεία που θα ακολουθήσουν τα ζητήματα της ισότητας. Η δύσκολη κατάσταση της πραγματικής οικονομίας, οι σοβαροί περιορισμοί των δημοσίων οικονομικών επηρεάζουν τις γυναίκες. Ένα μεγάλο ποσοστό γυναικών εργάζεται είτε με καθεστώς μερικής απασχόλησης, είτε με συμβόλαια περιορισμένης διάρκειας, προκειμένου να εξορροπήσουν την επαγγελματική με την οικογενειακή ζωή σε περιόδους οικονομικής κρίσης οι γυναίκες είναι πιο ευάλωτες. Μπροστά σε αυτές τις δυσκολίες είναι απαραίτητο να τοποθετήσουμε στο κέντρο των πολιτικών μας μια από τις βασικές αρχές της συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την αρχή της πλήρους και ουσιαστικής ισότητας ανδρών και γυναικών. Η επένδυση στην ισότητα είναι απαραίτητη και για την επίτευξη δικαιοσύνης και απόδοσης των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, αλλά και για να καταστήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση μια ένωση ανταγωνιστική και καινοτόμα. Είναι γεγονός ότι η θέση της γυναίκας έχει αναβαθμιστεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Υπήρξε σημαντική πρόοδος στην πρόσβαση και πρόθεση των γυναικών στην αγορά εργασίας, τα μορφωτικά επίπεδα των γυναικών τείνουν να είναι ψηλότερα από αυτά των ανδρών και ο ευρύτερος ρόλος τους στην οικονομία, στην κοινωνία και στην πολιτική αναβαθμίζεται. Εν τούτης, είμαστε ακόμη πολύ μακριά από τον στόχο της πλήρους ισότητας. Οι διακρίσεις είναι ακόμα ορατές σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένης και της απασχόλησης οι γυναίκες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα στην πρόσβαση και παραμονή τους στην αγορά εργασίας. Τα ποσοστά χάσματος αμοιβών και διαχωρισμού στην αγορά εργασίας εξακολουθούν να είναι ψηλά. Η συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική ζωή και στα κέντρα λήψης αποφάσεων είναι σε χαμηλά επίπεδα. Οι γυναίκες απομίζονται το μεγαλύτερο βάρος των οικογενειακών υποχρεώσεων και η μερική και η προσωρινή απασχόληση είναι πιο συνήθιση στις γυναίκες με αποτέλεσμα να διατρέχουν ψηλό κίνδυνο περιθωριοποίησης σε επισφαλείς δουλειές, με χαμηλό μισθό, δυσμενείς εργασιακές συνθήκες και ανεπαρκή συνταξιδοτικά δικαιώματα, ενώ τα φαινόμενα της βίας, της εμπορίας και της διακίνησης ανθρώπων επηρεάζουν κατά κύριο λόγο τις γυναίκες. Το νομοθετικό πλαίσιο στον τομέα της ισότητας έχει συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη του στόχου της ισότητας. Σε αυτή τη διαδικασία καθοριστική ήταν η συμβολή των πρωτοβουλειών και οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και ο ρόλος του Ευρωκοινοβουλίου. Από μόνη της όμως η νομοθετική κατοχήρωση της ισότητας δεν είναι αρκετή αν δεν μεταφράσουμε τους νόμους σε πράξη. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για κάθε κράτος μέλος να διασφαλίσει την εφαρμογή της νομοθεσίας και να θέσει σε ισχύ αποτελεσματικούς μηχανισμούς παρακολούθησης της εφαρμογής της. Ταυτόχρονα, η ουσιαστική ισότητα προϋποθέτει μεταξύ άλλων αλλαγή των στερεοτύπων και την αντιλήψεων, θέσπιση σωστών βάσεων από την παιδική ηλικία, ενσωμάτωση της αρχής της ισότητας σε όλο το οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθε. Βασική επιδίωξη της Κυπριακής Προεδρίας είναι να εργαστεί προς την κατεύθυνση μιας καλύτερης Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτού του κεντρικού μηνύματος, η Κυπριακή Προεδρία επιθυμεί να συνεισφέρει στην πρόθεση βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. μια ανάπτυξης που να βασίζεται στις αρχές της αλληλεγγύης και με κύριο προσανατολισμό την παροχή ενός καλύτερου μέλλοντος για τις νέες γενιές αλλά και για όλους τους πολίτες της Ένωσης, άνδρες και γυναίκες. Έχετε ήδη ενημερωθεί από τον συνάδελφο μου Υπουργό Δικαιοσύνη και Δημόσια Τάξη για κάποια από τα θέματα στα οποία θα επικεντρωθεί η Προεδρία σε σχέση με τα θέματα. Θα ήθελα να επισημάνω και εγώ με τη σειρά μου τη σημασία που δίνουμε στην πρόληψη και την καταπολέμηση όλων των μορφών βία ενάντια στι γυναίκε. Πολλέ φορέ τείνουμε να επικεντρωνόμαστε σε θέματα που σχετίζονται με την ισότητα στην απασχόληση και αυτό είναι σωστό γιατί η απασχόληση και η πρόσβαση στην εργασία είναι βασικό κριτήριο για την ισότητα. Ωστόσο, το γεγονός ότι η βία εξακολουθεί να πλήττει ένα μεγάλο αριθμό γυναικών είναι απαράδεκτο. Είναι εξαιρετικά σημαντικό για την Κυπριακή Προεδρία να επαναφέρουμε το θέμα αυτό στο προσκήνιο και να συμβάλλουμε στην αποτελεσματική καταπολέμηση του φαινομένου. Είναι γι' αυτό το λόγο άλλωστε που έχουμε επιλέξει να ασχοληθούμε με τους δείχτες της πλατφόρμας του Πεκίνου, οι οποίοι καταπιάνονται με το θέμα αυτό και ειδικότερα με τα θέματα υπηρεσιών στήριξη θυμάτων. Κύριος μας στόχος είναι να υιοθετηθούν συμπεράσματα του Συμβουλίου για το θέμα και να αξιοποιηθεί όσο το δυνατόν καλύτερα η σχετική μελέτη για το θέμα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα Φύλων. Μεταξύ των προτεραιοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας περιλαμβάνεται και το ζήτημα της ευζοίας και της καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού των παιδιών. Για το θέμα αυτό θα επιδιωχθεί η υιοθέτηση συμπερασμάτων του Συμβουλίου. Στόχος είναι όπως μεταξύ των θεμάτων που θα εξεταστούν να περιληφθεί και το θέμα της στήριξης της απασχόλησης για οικογένειες με παιδιά μια απαραίτητη προϋπόθεση για να καταπολεμήσουμε, τη φτώχεια ανάμεσα στα ίδια τα παιδιά. Σημειώνω ότι για αυτή την προτεραιότητα έχει προγραμματιστεί συνέδριο Προεδρίας τον Οκτώβριο του 2012, στο οποίο θα κληθεί να συμμετάσχει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μια ακόμη σημαντική προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας στον τομέα της ισότητας σχετίζεται με το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Έχουμε ιδιαίτερη ευαισθησία στο θέμα, μιας και η Κύπρος συγκαταλέγεται στα κράτη-μέλη με ψηλό χάσμα αμοιβών, 21% περίπου. Οι αιτίε του χάσματος είναι αναφίβολα πολλέ. Η απασχόληση μεγάλου ποσοστού γυναικών σε ανειδίκευτα επαγγέλματα και σε χαμηλά αμοιβόμενου τομεί οικονομική δραστηριότητα είναι μια από τι αιτίε. Από την άλλη, το φαινόμενο του μισθολογικού χάσματο παρατηρείται και σε επαγγελματικέ δραστηριότητε ψηλότερη ειδίκευση. Κάτι που καταδεικνύει ότι οι διαφορέ στι αμοιβέ μεταξύ των φύλων δεν εξαλείφονται ούτε όταν οι γυναίκε ανελίσσονται στι ψηλότερε βαθμίδε τη ιεραρχία, αναγνωρίζοντα τη σημασία που έχει η περαιτέρω διαρεύνηση αυτού του θέματο και η συνέχιση τη προσπάθεια για εξέβρεση λύσεων με στόχο την οριστική εξάλληψη αυτού του φαινομένου, η Κυπριακή Προεδρία έχει θέσει υπό την αιγίδα της τριμερές συνέδριο για το χάσμα αμοιβών. Στο συνέδριο τα κράτη-μέλη θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν τις διάφορες προκλήσεις αλλά και να προσδιορίσουν καλές πρακτικές πάνω στο θέμα. Ένας από τους στόχους είναι να αναδειχτούν πρακτικές και μέτρα που μπορούν να εφαρμοστούν από τις ίδιες τις επιχειρήσεις προκειμένου να εξαλειφθεί το χάσμα αμοιβών και να προωθηθεί η αρχή της ισότητας μεταξύ των δύο φύλων. Θέλω να υπογραμμίσω ότι για τη θεματολογία του συνεδρίου έχουμε μελετήσει και αξιοποιούμε την πραγματικά αξιόλογη έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφορικά με τις συστάσεις προς την Επιτροπή για την εφαρμογή της αρχής της ισομισθίας. Και αναφίβολα το Ευρωκοινοβούλιο θα είναι ένας από τους προσκεκλημένους μας για να δώσει τη δική του συμβολή σε αυτό το συνέδριο. Σε ό,τι αφορά την οδηγία και την προστασία των εγγύων εργαζομένων, λεχών και γαλουχωσών εργαζομένων, παρά τις δυσκολίες, εξακολουθούμε να πιστεύουμε και ότι υπάρχει η ανάγκη, αλλά υπάρχει και η πρόθεση από την πλευρά της Κυπριακής Προεδρίας να εργαστούμε για να εξεύρουμε μια ισορροπημένη λύση. Μια λύση που θα είναι προς το συμφέρον της μητέρας και του παιδιού, αλλά και της οικογένειας ως σύνολο. Προς το σκοπό αυτό έχουμε κάθε καλή διάθεση να εργαστούμε τόσο εντός του Συμβουλίου αλλά και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με στόχο να βρούμε τις κοινέ συνισταμένες που θα, μας θα μας επιτρέψουν να προχωρήσουμε αυτό το σημαντικό κεφάλαιο. Πρόσθετα, η Προεδρία θα συνεχίσει την εργασία σε σχέση με την ολοκλήρωση του νομοθετικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση συνεχίζοντας στη βάση της εργασίας που έκαναν η Πολωνική και η Δανική Προεδρία σε σχέση με τους πρόνοιες που αφορούν την ηλικία ως παράγοντα διάκρισης, αφού και η γενική διαπίστωση του Συμβουλίου είναι ότι οι εν λόγω πρόνοιες χρήζουν περαιτέρω εξέτασης. Θα ήθελα να καταλήξω επαναλαμβάνοντας ότι προσβλέπουμε στη στενή και επικοδομητική συνεργασία σας για να προωθήσουμε εκείνες τις πολιτικές που θα βοηθήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να ανακάμψει σε συνθήκες ανάπτυξη με κεντρικό στόχο την ευημερία και τη διασφάλιση ψηλού επίπεδου ποιότητας ζωής για τον κάθε πολίτη της Ένωσης. Είμαστε πάντοτε πρόθυμοι στα πλαίσια ενός ειλικρινούς και ανοιχτού διαλόγου με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μεταφέρουμε τις θέσεις του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και να εργαστούμε ως Προεδρία για να εξεύρουμε ισορροπημένες κοινά αποδεκτές λύσεις. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας δίνετε και εύχομαι καλές διακοπές σε όλους. Σας ευχαριστώ πολύ. κυρία και κύριε Υπουργέ, κυρία Χαραλάβους, κύριε Λουκά, για τις παρουσιάσεις σας. Σας διαβεβαιώ ότι δεν είμαι ο μόνος εδώ μέσα που περιμένει με αδημονία τις διακοπές και τη θερινή ραστόνη. Ίσως εσείς χρειάζεστε μια πρώτη ανάπαυση πριν αρχίσουν, ε, αρχίσει η σκληρή δουλειά από Σεπτέμβριο ίσως. Πάντως ευχαριστώ πολύ για τα πολύ καλά σας λόγια. Επιβεβαιώνετε ε, με τα λόγια σας, τα όσα είδαμε εμείς οι στην επίσκεψη στην Κύπρο, ότι δηλαδή ε, υποστηρίζετε διακαώς την ε, ισότητα των φύλων, ότι έχετε θέσει το θέμα αυτό πολύ ψηλά στην ημερησία διάταξη και ότι θα προωθήσετε όλα τα ζητήματα. Φυσικά είμαστε ευγνώμονες για αυτή την προσοχή που δίνετε στα θέματα της ισότητας των φύλων. Εμείς ιδιαίτερα από την Επιτροπή μας θα είμαι βεβαίως παρόν στη διάσκεψη που θα οργανώσετε για το θέμα της βίας της βάρος των γυναικών προσωπικώς εγώ το φθινόπωρο. Ε, τώρα θα απευθύνω το λόγο στους συντονιστές μας στις και τους συντονιστές, εάν θέλει κάποιος να λάβει το λόγο και να υποβάλει ερωτήσεις. Στη συνέχεια μπορούν να απαντήσουν οι υπουργοί και σε ένα δεύτερο γύρο ερωτήσεων τα λοιπά μέλη της Επιτροπής μας μπορούν να διατυπώσουν ερωτήσεις πάλι με την απάντηση εκ μέρου της κυρίας και του κυρίου Υπουργού. Έχουμε στην Επιτροπή μας, ξέρετε, πολύ δραστήρια μέλη, στρατευμένα μέλη. Έχουμε συναδέλφους ε, που περιμένουν με αδημονία να μιλήσουν, να εκφράσουν τις απόψεις τους και γι' αυτό το λόγο είμαι υποχρεωμένο να ορίσω χρονικά όρια στις ερωτήσεις των βουλευτών για να έχουμε αρκετό χρόνο να ακούσουμε τις απαντήσεις των ε, δύο υπουργών μας σήμερα. Ανάλογα λοιπόν και με την εκπροσώπηση των πολιτικών ομάδων στην Επιτροπή μας, αν και βλέπω ότι δεν έχουμε το συντονιστή εκ μέρους του ΕΛΚ εδώ σήμερα, ε, άρα θα, θα τον ακούσουμε αργότερα. Και έτσι ξεκινώ με την κυρία Τόμσον για τρία λεπτά παρακαλώ. Eh. Ακούγεται η ελληνική καμπίνα, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Μα ακούτε, όχι, στο έφτα. Συγγνώμη, κάποιο λάθο υπήρχε με τα κοπιά. Σα ευχαριστώ λοιπόν και πρέπει να πω ότι είναι πολύ εντυπωσιακό και φιλόδοξο το πρόγραμμα που έχετε ορίσει. Έχετε θέσει το δάκτυλο επί τον τύπο των ύλων στα κύρια θέματα που πρέπει να μας απασχολήσουν ως προς την ισότητα των φίλων. Καταρχάς, αυτό που είπατε για την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και την καταπολέμηση των ε, διακρίσεων της βάρος των γυναικών στην αγορά εργασίας είναι πάρα πολύ σημαντικά για την ανταγωνιστικότητα μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως, Εάν κοιτάξουμε και την ουσία του θέματος, τα πιο βασικά πράγματα δηλαδή, το θέμα της βίας των γυναικών είναι πάρα πολύ σημαντικό, ένας αγώνας τον οποίο θα πρέπει διαρκώς να αποδιόμαστε όλοι μαζί και πρέπει να περιορίσουμε σημαντικά αυτό το φαινόμενο το οποίο είναι πολύ εκτεταμένο σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι κάποια κράτη-μέλη γνωρίζουν περισσότερη βία από ό,τι άλλα. Είναι ένα θέμα που πρέπει να συζητήσουμε, είναι ένα θέμα στο οποίο πρέπει να λάβουμε δράση. Επίσης, το θέμα της κοινωνικής πρόνοιας. Εγώ σοσιαλίστρια ιδιαίτερος θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό το θέμα της κοινωνικής πρόνοιας, πρέπει να το φροντίσουμε. Είναι ένας τρόπος να καταπολεμηθεί η φτώχεια. Ε, η διαφορά στις αμοιβέ είναι επίσης σημαντική και εδώ ξέρετε έχετε πρωτοπορία διότι έχουμε ήδη μία έκθεση εμείς στην Επιτροπή μας για την διαφορά στις αμοιβέ Θέλουμε να επανεστιαστούμε στο θέμα αυτό. Είχαμε μια πρώτη έκθεση το 2006 ως προς τις ε, διαφορές ε, αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Δεν έχει φέρει τους αναμενόμενους καρπούς. Υπάρχουν ακόμη σημαντικά προβλήματα και ανισότητα στις αμοιβέ και έτσι θέλουμε να αναθεωρηθεί η οδηγία. Θέλουμε να ξανανοίξει δηλαδή το ε, θέμα της ισχύουσας νομοθεσίας έχοντας υπόψη όλη τη νέα γνώση και τον τρόπο που μπορούμε να καταπολεμήσουμε τις διαφορές στην αμοιβή ε, είμαι πολύ ευτυχής λοιπόν και περιμένω και εγώ να πω ότι θα έρθει η ώρα να γίνει αυτή η διάσκεψη. Δεν ξέρω αν έχετε συγκεκριμένα στοιχεία για τις ημέρες που θα οργανωθεί αυτό ε, να μας ενημερώσετε γιατί ξέρετε έχουμε πολύ πιεσμένο πρόγραμμα και θέλουμε να οργανωθούμε. Ταυτόχρονα πάντως θέλω να σας συγχαρώ ήδη από τώρα για την ε, οδηγία, για την πρωτοβουλία για την οδηγία για την άδεια μητρότητας και της ε, μητέρας όταν θυλάζουν ε, το μωρό τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Κυρία λεπτά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Θα ήθελα καταρχάς να συγχαρώ τους εκπροσώπους της Κυπριακής Προεδρίας για το ιδιαίτερα φιλόδοξο πρόγραμμά τους. Ένα ευαίσθητο ζήτημα για την δική μας την Επιτροπή είναι η βία κατά των γυναικών. Ήδη από την αρχή της θητείας έχουμε προσπαθήσει να καταπολεμήσουμε το ζήτημα αυτό χωρίς συγκεκριμένα αποτελέσματα. Είπατε ότι δεσμεύεστε πάρα πολύ για τη στρατηγική της καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών. Για μας το ζήτημα είναι πώς θα γίνει κάτι τέτοιο. Πώς μπορείτε να επιταχύνετε, να κινητοποιήσετε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς επίσης και τα κράτη-μέλη για το ζήτημα αυτό. Και έχετε δεσμευθεί, όπως είπατε, να καθορίσετε το 2015 ως έτος, ευρωπαϊκό έτος για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Τι προβλέπετε να κάνετε σε σχέση με αυτό συγκεκριμένα. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι είχαμε μια πολύ επικοδομητική συνεργασία με την Δανέζικη Προεδρία όσον αφορά το ζήτημα της βίας κατά των γυναικών και καταφέραμε να έχουμε πολύ θετικές διαπραγματεύσεις όσον αφορά μια οδηγία για την προστασία των θυμάτων εγκληματικών πράξεων. Φαντάζομαι ότι αυτό θα επιβεβαιωθεί και από την Επιτροπή μας σήμερα το απόγευμα. Θα έχουμε πάντως και τις διαπραγματεύσεις στα πλαίσια του EPO, του Ευρωπαϊκού Διατάγματος Προστασίας και στα πλαίσια της Κυπριακής Προεδρίας. Ως προς αυτό, πώς θα συνεργαστείτε με τα κράτη-μέλη, έχετε ήδη κάποιες πρώτες πληροφορίες από τα κράτη-μέλη. Και μια τελευταία ερώτηση την Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Σε σχέση με τη σύμβαση αυτή μπορείτε πάλι ή έχετε κάποια σχέδια για να κινητοποιήσετε τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να υπογράψουν τη σύμβαση αυτή και να έχουμε μια ισχυρή θέση ως Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια αυτής της σύμβασης. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Κορνέλη, για δυόμιση λεπτά. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη, γιατί πρέπει δυστυχώς να αποχωρήσω από την αίθουσα για να ψηφίσω σε μια άλλη κοινοβουλευτική επιτροπή. Ξέρετε ότι είναι η τελευταία εβδομάδα πριν τις θερινές διακοπές και προσπαθούμε όλοι οι ευρωβουλευτές να πληρώσουμε τις αρμοδιότητές μας σε διάφορες κοινοβουλευτικές επιτροπές. Θα είμαι λοιπόν πολύ σύντομη. Αναφερθήκατε στη στρατηγική Ευρώπη 2020. Είχα την ιδιαίτερη χαρά να μιλήσω με την κυρία Χαραλάμπους και στο παρελθόν και μου είχε πει ότι θα αναφερόταν στο ζήτημα της δημοκρατίας καθώς επίσης και της συμμετοχής των συμβαλωμένων ενδιαφερομένων μερών στο, στα πλαίσια του εξαμήνου. Τι ακριβώς πρόκειται να γίνει με το ζήτημα της συμμετοχής ε, των γυναικών στα πλαίσια της στρατηγικής αυτής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ζήτημα του gender mainstreaming να ληφθεί υπόψη στα πλαίσια της στρατηγικής ε, αυτής γιατί αυτό θα πειράσει πάρα πολύ και το ζήτημα της απασχόλησης, καθώς επίσης και το ζήτημα της καταπολέμησης της φτώχειας. Ξέρετε ότι είναι κυρίως οι γυναίκες αυτές οι οποίες πλήττονται από το φαινόμενο της φτώχειας. Υπάρχουν επίσης κάποια εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα, τα οποία περιλαμβάνουν τη διάσταση του φύλου, αλλά πάλι εθνικά προγράμματα δεν περιλαμβάνουν καθόλου τη διάσταση του φύλου. Θα ήταν λοιπόν πολύ σημαντικό να δούμε στα πλαίσια του εξαμήνου αυτού τι θα γίνει με αυτές τις χώρες, αν γίνεται τουλάχιστον να, γίνει μια συζήτηση στα πλαίσια του Συμβουλίου, προκειμένου όλα τα κράτη-μέλη να συμφωνήσουν για το ζήτημα της ε, συμμετοχής των φύλων. Ε, ε, e Η κυρία Κράτσα, δεν το είχα συνειδητοποιήσει ότι αντικαθιστά το συντονιστή του ΕΛΚ. Έχετε το λόγο κυρία Κράτσα για τρία λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους εκπροσώπους, τον κύριο Υπουργό, την κυρία Υπουργό, τους εκπροσώπους της Κυπριακής Κυβέρνησης και της Κυπριακής Προεδρίας σε αυτή την ανταλλαγή απόψεων σήμερα με την Επιτροπή μας. Είναι πολύ σημαντικό για μας ότι είναι μία από τις προτεραιότητάς σας η ισότητα των φύλων και πολύ καλά το τοποθετήσατε από την πλευρά των αξιών και των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και από την πλευρά της ε, ανάπτυξης ε, μιας οικονομίας με ευημερία και συνοχή. Ε, ήθελα να, να ε, σημειώσω τρία πράγματα. <clears throat> Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μας ότι ε, το θέμα της συμμετοχής των γυναικών στις αποφάσεις των οικονομικών φορέων και πιο συγκεκριμένα στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων είναι στις προτεραιότητές σας αναφέρθηκε διεξοδικά ο Υπουργός. Έχω όμως μια απορία πώς δεν ε, αναφέρεστε στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συγκεκριμένα είμαι η συγγήτρια αυτής της έκθεσης, η οποία παρουσιάζει το πρόβλημα αυτό την, ε, και προτείνει μια στρατηγική επίτευξη αυτού του στόχου, στρατηγική η οποία δεν έχει μόνο να κάνει με την ε, ανάγκη υιοθέτηση δεσμευτικών μέτρων, για την συμμετοχή των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια, αλλά και μια ευρύτερη στρατηγική ε, αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού που θα δώσει την ευκαιρία να, έρχονται, να φτάνουν οι γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια χωρίς να χρειάζονται ε, άμεσες παρεμβάσεις όπως είναι αυτή των δεσμευτικών μέτρων. Ε, είμαι έκπληκτη λοιπόν πώς δεν, δεν έχετε ενημερωθεί για τη θέση του Κοινοβουλίου και τις απαιτήσει που εκφράζει το Κοινοβούλιο τόσο στην Κομισιόν όσο και στο Συμβούλιο. Και δεύτερον, δεν κατάλαβα κύριε Υπουργέ, ποια στο θέμα αυτό είναι η δική σας θέση. Μας είπατε ότι υπάρχουν κράτη τα οποία στη, ζητούν δεσμευτικές ε, παρεμβάσεις, υπάρχουν κράτη τα οποία, κύριε Υπουργέ, ήδη έχουν υιοθετήσει δεσμευτικές παρεμβάσεις, υπάρχουν άλλα κράτη τα οποία θέλουν να δώσουν ακόμη περιθώριο στις κυβερνήσεις δεν ξέρουμε ποια θα είναι θέση της Κυπριακής Προεδρίας. Είναι πολύ σημαντικό για μας, διότι πέρυσι τον Ιούλιο ψηφίστηκε η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ζητούσε σε ένα χρόνο, δηλαδή σήμερα, από την Επιτροπή να, πάρει δεσμευτικές, ε, ε, να κάνει δεσμευτικές παρεμβάσεις αν δεν έχει επέλθει πρόοδο. Ναι. Επειδή πρόοδο δεν έχει επέλθει, ήρθε η ώρα να, κάνουμε, να ανανεώσουμε την έκκλησή μα τόσο στο Συμβούλιο όσο και στην Επιτροπή. Ε, είναι λοιπόν σημαντικό για μας να μάθουμε τη δική σας θέση. Το άλλο θέμα. Ε, ασχοληθήκατε με τις αδικίες και με τις ανισότητες που ήδη υπάρχουν και τις πρωτοβουλίες της δικές σας. Ε, εγώ ήθελα να σας ζητήσω εκ μέρους της πολιτικής μου ομάδας ποια στρατηγική μπορείτε να εφαρμόσετε για να δούμε την εφαρμογή του δικαίου που ήδη έχουμε. Η Ευρώπη έχει ένα υψηλό πλωστάσιο δικαίου. Η Επιτροπή μας ήταν πρόσφατα στις Ηνωμένε Πολιτείε, για να μην αναφερθώ για άλλες περιοχές του κόσμου. Αναφέρομαι στο μοντέλο το δυτικό, το, άλλο μοντέλο το δυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών και ε, είδαμε, διαπιστώσαμε η διεισόμαση την υπεροχή που έχει το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο και στον τομέα αυτό της ισότητας. Πρέπει λοιπόν, έχουμε ανάγκη από μια Προεδρία με ευαισθησία όπως εσείς, να κάνει πράγματι να ε, ζητήσει μια ε, απογραφή της μη εφαρμογής του νόμου. Συμφωνώ μαζί σας ότι είμαστε σε μια πολύ ευαίσθητη φάση, εποχή κρίση οικονομικής και δεν πρέπει να παραμελήσουμε το κοινωνικό μοντέλο στο στόχο της επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων, διότι συμφωνούμε μαζί σας ότι η ισότητα αντίθετα θα δώσει ε, ε, έναυσμα ανάπτυξης και κίνητρα ανάπτυξης στην κοινωνία μας και στην οικονομία μας, άρα και επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων. Κλείνοντας, είναι η άλλη παρατήρηση εκ μέρους της πολιτικής μας ομάδας. Θέλουμε ε, να προβάλλουμε τα θετικά μοντέλα της επίτευξης ε, των, επιτεύξεων των κοινωνικών στόχων ε, από τις ε, Ευρωπαίες γυναίκες. παράλληλα με τις ανισότητες, παράλληλα με τις διακρίσεις που πρέπει ακόμη να καταπολεμήσουμε, πρέπει να αναδείξουμε, ιδίως στην εποχή αυτή που υπάρχει απεσιοδοξία στην ευρωπαϊκή οικονομία και κοινωνία, το θετικό ρόλο και τα θετικά μοντέλα των Ευρωπαίων γυναικών που διαπρέπουν σε πολλούς τομείς. Όχι μόνο της πολιτικής και της οικονομίας, αλλά οι γυναίκες μεγάλες καλλιτέχνες που δίνουν μεγάλη ακτινοβολία στις χώρες του και στην Ευρώπη, μεγάλες ερευνήτριες, κατακτήσει σε όλο τον κόσμο. Και θέλω να σας ζητήσουμε να πάρετε μια πρωτοβουλία για να προβληθεί αυτή η θετική εικόνα ανά τον κόσμο των Ευρωπαίων γυναικών. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Με συγχωρείτε, δεν γνώριζα ότι αντικαθιστάτε το συντονιστή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο. Τώρα είμαι ενήμορο. Και επαναρχόμαστε τώρα στον κατάλογο των ομιλητών, η κυρία Γιάννα Κουδάκη. Ε, ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι πολύ σύντομη γιατί πρέπει και εγώ να φύγω σε μια συνεδρία. Θα θέλω να καλωσορίσω την Κυπριακή Προεδρία. Περίμενα με αδημονία να ξεκινήσει. Άκουσα τα σχόλια των Υπουργών που ωστόσο πρέπει να σας πω ότι κάπως με στεναχωρούν ως Βρετανή βουλευτή γιατί έχει δίκιο ο Πρόεδρος. Είμαστε ενωμένοι, είμαστε μια ομάδα στην ε, Επιτροπή των Γυναικών και αγωνιζόμαστε για το καλό των γυναικών στους διάφορους τομείς η ομάδα μας των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών, όπως ίσως γνωρίζετε, αισθάνεται ανησυχία για τα σχόλια που κάνατε ως προς την άδεια μητρότητας. Πολύ φοβούμαι ότι μπαίνετε σε μία σύραγγα η οποία δεν θα σας οδηγήσει στην επιτυχία όπως θα το επιθυμούσατε ίσως. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ως προς το θέμα της απασχόλησης γιατί ανήκει τα αρμόδια των κρατών μελών και εγώ θα προτιμούσα να ε, προχωρήσουμε περισσότερο προς μια επιλογή ανταλλαγής βέλτιστων των πρακτικών και χειραφέτησης των γυναικών. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ρωτήσω αν έχετε κάτι στο πρόγραμμά σας για την ε, χειραφέτηση των γυναικών, για την ενίσχυση της παρουσίας τους, αλλά όχι νομοθετικά την ε, ενίσχυση των δυνατοτήτων του να διεκδικήσουν θέσει υψηλέ σε διοικητικά συμβούλια και το Και για το θέμα βέβαια τη βία βάρο των γυναικών, ένα ζήτημα το οποίο μα απασχολεί ιδιαίτερω. Εγώ είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ και πρόσφυγε από την Κύπρο και έτσι γνωρίζω αρκετά τα, τα θέματα αυτά. Ένα ζήτημα στο οποίο δεν αναφερθήκατε και με καταπλήσει αυτό είναι το θέμα της διακίνησης που λαμβάνει χώρα από ό,τι γνωρίζω και στην Κύπρο. Μπορείτε να μα δώσετε τις απόψεις για, ε, για το θέμα τη διακύπνηση ανθρώπων. Για δε τη χειραφέτηση θα ήθελα πιο πολλά στοιχεία ε, ως προς το πώς βλέπετε το θέμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και πώς μπορείτε να κινητοποιήσετε περισσότερε γυναίκες ώστε να αναλάβουν δραστηριότητα, να ε, θέσουν ε, να ιδρύσουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις τα λοιπά. Ε, δυστυχώς πρέπει να φύγω, αλλά ο βοηθός μου εδώ θα αναλάβει να κρατήσει σημειώσεις για τις απαντήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Ζούμπερ. Πρόεδρε, η κυρία, κυρία Γκουρμάη, με συγχωρείτε. Η κυρία Ζούμπερ προηγείται. Obrigada, Sr. Presidente. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω την Κυπριακή Προεδρία και τους δύο υπουργούς. η συνάντηση της, η επίσκεψη αυτής της Επιτροπής στην Κύπρο ήταν πραγματικά πολύ ωφέλιμη και επικοδομητική. Μας επέτρεψε να ανταλλάξουμε απόψεις και να ενημερώσουμε για τις ανησυχίες μας. Μας υποδεχτήκατε πολύ ευγενικά και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γι' αυτό. Ε, θα ήθελα να σας αναφέρω ορισμένε μας ανησυχίες και εδώ, γιατί ζούμε μια εποχή πολύ περίπλοκη και ανησυχητική για το ε, θέμα της ε, πολιτιστικής προόδου που είχαν καταφέρει οι γυναίκες τα τελευταία χρόνια σε θέματα ισότητας. Αυτό το θέμα δεν μπορούμε να το δούμε αποκομμένο. Δηλαδή, από τη μια μεριά οι γυναίκες και από την άλλη μεριά οι κοινωνικές και οι οικονομικές πολιτικές. Αυτά τα δύο θέματα συνδέονται. Θα πρέπει να τα δούμε από κοινού. Κατά την άποψή μας, όλη η πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δίνει μια μείωση της παρέμβασης του κράτους και μια μείωση των δικαιωμάτων. Αυτό έχει επηρεάσει πάρα πολύ τα δικαιώματα των γυναικών. Ιδιαίτερα των γυναικών των λαϊκών στρωμάτων, των εργαζόμενων γυναικών οι οποίες ε, έχουν εντυπωσιακά ποσοστά φτώχειας πλέον. Τέσσερα θέματα θέλω να θέσω. Πρώτον, η ανεργία. Προφανώς είναι ανησυχητικό γενικά, αλλά ειδικά για τις γυναίκες είναι ακόμα χειρότερο. Όχι μόνο λόγω της αύξησης της ανεργίας, αλλά και για το όσα αυτό σημαίνει σε ό,τι αφορά την ε, αδυναμία ε, διατήρησης της ανεξαρτησίας τους. επιστρέφουμε σε μια πορεία ανισότητα στην οποία πιστεύαμε ότι είχαμε αφήσει πίσω. Απ' την άλλη μεριά έχουμε το θέμα των νέων μορφών εργασίας. Το πακέτο απασχόλησης που θα προτείνει η Κομισιόν δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ευελιξία στην αγορά εργασίας. Αυτή η ευελιξία θα φέρει υποτίθεται μια οικονομία πιο ανταγωνιστική και η Κομισιόν δίνει ιδιαίτερη σημασία στις πιο επισφαλείς θέσεις εργασίας, τα στάζ και τα σεμινάρια μαθη... της περίοδου μαθητείας και λοιπά. Κάτι που για μας είναι ε, θέσεις εργασίας ε, πραγματικά επισφαλείς και καθόλου σταθερές. Και οι γυναίκες πλέονται πιο πολύ από όλους από τέτοιου είδους θέσεις Αυτέ οι σχέσεις εργασία οι ασταθείς, έχουν όμως και άλλες επιπτώσεις για τις γυναίκες. Γιατί πολύ συχνά μιλάμε για την κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική συμμετοχή των γυναικών. Όμω, πέραν αυτών, στην πράξη, αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβάλλει μια πλήρη απορρίθμιση της ζωής της γυναίκας, αυτό Προφανώ της αφαιρεί δυνατότητε να συμμετάσχει στην κοινωνία. Δηλαδή είναι μια γυναίκα, δουλεύει σε μια επιχείρηση και δεν ξέρει πού θα δουλεύει την επόμενη εβδομάδα, πότε θα δουλεύει την επόμενη εβδομάδα, τι ωράρια κλπ. Και δεν μπορεί να το διαπραγματευτεί, είναι προφανέ ότι θα πληγεί η δυνατότητά τη να συμμετάσχει στην κοινωνία. Υπάρχουν δύο-τρία άλλα θέματα, ε, επίσης που είναι σημαντικά να το σκεφτούμε. Πρέπει να δούμε αν υπάρχει ένα καινούριο φαινόμενο πρώτον στο πλαίσιο της ενδοοικογενειακής βίας που έχει σχέση με την κοινωνική και οικογενειακή σταθερότητα και δεύτερον το κατά πόσον έχει αυξηθεί η πορνεία ε, ως αποτέλεσμα της δραματικής κατάστασης που ζουν πολλές γυναίκες. Να δούμε δηλαδή αν η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει την ενδοοικογενειακή βία και την πορνεία. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να, το, να, να μας προβληματίσει. Και πρέπει να δούμε όλα, όλες τις τυχές, όχι μόνο μία ή δύο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν νομίζω ότι από την ομάδα EFD θέλει κανείς το λόγο ή από τους μη εγγεγραμμένους. Επομένως, θα απευθυνθώ και πάλι στους υπουργού προκειμένου να δώσουν σύντομες απαντήσεις στις ερωτήσεις που ακούστηκαν και θα έχουμε και ένα νέο γύρο ερωτήσεων από άλλους βουλευτές που έχουν ζητήσει και αυτή το λόγο. Μία ερώτηση ακόμα. Δεν συμφωνείτε, κύριε Τρόλε, με αυτό. Λοιπόν, θα κάνουμε το εξή. Θα ακούσουμε ακόμα κάποιες ερωτήσεις και, τότε, και στη συνέχεια μόνο θα δώσουμε το λόγο στους υπουργού. Για δύο λεπτά λοιπόν, η κυρία Γκουρμάη και η κυρία Γερακόφ στη συνέχεια. Κυρία Γκουρμάη, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους Υπουργούς για την πολύ σημαντική τους συνδρομή, καθώς και για τόσα μας είπαν για την Κυπριακή Προεδρία, όσον αφορά ιδίω το ζήτημα της κοινωνικής ευαισθησίας και της αλληλεγγύης. Θα πρέπει να προωθήσουμε τις προτεραιότητες αυτές, ιδίω όταν διανύουμε μια περίοδο οικονομικής κρίσης. Χρειαζόμαστε επίσης μια ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμού στα πλαίσια της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν ενσωματωθεί διάσταση του φύλου. Οι γυναίκες ε, είναι από τις πιο ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας, που μένως θα πρέπει να κινητοποιηθούν όλα τα απαραίτητα μέσα στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό επίση να ασχοληθούμε με το ζήτημα τη βία κατά των γυναικών. Μιλήσατε εκτενώ και οι δύο για το ζήτημα αυτό και πολύ θετικά. Και όντω το 2015 θα μπορούσε να κηρυχθεί ω Ευρωπαϊκό Έτο τη καταπολέμηση τη βία κατά των γυναικών. Είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό για μα. Χαιρετίζουμε επίση τη δέσμευση τη Κυπριακή Προεδρία όσον αφορά το ζήτημα του μισθολογικού χάσματο. Όντω και εμεί, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχουμε ασχοληθεί εντόνω με το ζήτημα αυτό. Βέβαια, δεν αρκούν κάποιε δεσμεύσει θεωρητικέ. Χρειαζόμαστε μια πραγματική δέσμευση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συμμετοχή επίση των γυναικών στην κοινωνική ζωή, η κυρία Κράτσα αναφέρθηκε εκτενώ στο ζήτημα αυτό. Η κυρία Ρέντινγκ, η Επίτροπος, θα μας πει επίσης τι έγινε στα πλαίσια της διαβούλευσης, ιδίως όσον αφορά την συμμετοχή των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των εταιριών. Θέλουμε επίσης να δούμε τι θα μπορούσε να γίνει μέχρι το 2015 ή το 2020 και να γνωρίσουμε από τώρα ποια είναι τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων. Η Κυπριακή Προεδρία έχει συγκεκριμένες προτεραιότητες και θα ασχοληθεί προφανώς και με το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020 και με τον προπολογισμό βέβαια για το 2013. Θα ήθελα λοιπόν να επιστήσω την προσοχή σας στο ότι χρειάζεται ένας προπολογισμό ο οποίος θα λαμβάνει υπόψη και το ζήτημα της ισότητας των φύλων και θα πρέπει επίση να ενσωματωθεί η διάσταση του φύλου τόσο στο πολιτέ νομοσυνομικό πλαίσιο, όσο όμω και στον προπολογισμό του 2013. Θα πρέπει σε όλα τα επίπεδα να υπάρχουν τα απαραίτητα κονδύλια για την πρόθεση των πολιτικών στι οποίε αναφερθήκατε και θα ήθελα επίση να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στην οδηγία και την προστασία των εγγύων εργαζομένων. Διάβασα επίση την επιστολή τη κυρία Ρέντινγκ και τη κυρία Βασιλείου αφορά του Ολυμπιακού Αγώνε Νομίζω πάντως ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταβληθούν ακόμα περισσότερες προσπάθειες όσον αφορά την εκπροσώπηση των γυναικών στον αθλητισμό και στους αρμοδίους, στις αρμόδιες αρχές για τον αθλητισμό. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ε, Γιάροκα, Κυρία Γιάροκα, έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομη. Η ερώτησή μου αφορά την φτώχεια των παιδιών ε, χαίρομαι ιδιαίτερως διότι, στην τριμερή κρατήσατε το θέμα της φτώχειας των παιδιών, οργανώνετε τη διάσκεψη, αλλά θα ήθελα πιο πολλά στοιχεία αν έχετε να μας δώσετε για το πώς προβλέπετε να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα αυτό. Αρκετές στρατηγικές αναπτύσσονται αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει στρατηγική για τους Ρωμά, υπάρχει στρατηγική για την αντιμετώπιση της κρίσης, που ίσως να είναι χρήσιμες για την Προεδρία σας και θα σας επιτρέψουν να προαγάγετε το θέμα αυτό ακόμη περισσότερο. Περιμένουμε βεβαίως ε, στην καλή συνεργασία μαζί σας στο θέμα της φτώχειας των παιδιών και να μας δώσετε κάποιες ιδέες για το τι περιμένετε να επιτύχετε στην, ε, στο εξάμεινό σας. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα θα ακούσω την κυρία Στρέλα, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τους ε, υπουργού για την παρουσίαση αυτού του φιλόδοξου προγράμματος. Ε, συμφωνώ με τις ε, προτεραιότητες που ανακοινώθηκαν, αλλά θα καταλάβετε προφανώς ότι ως εισηγήτρια της αναθεώρησης οδηγίας για την μητρική άδεια, θα πρέπει να εκφράσω την, ανησυχία, την ιδιαίτερη ανησυχία μου γιατί θα πρέπει το θέμα αυτό να ξεμπλοκαριστεί. Ε, τον Οκτώβριο του 2010 το Κοινοβούλιο ενέκρινε την ε, πρόταση αναθεώρησης αυτής της οδηγίας. Έχουν περάσει πλέον διάφορες προεδρίες, η Βελγική με την οποία συνεργαστήκαμε, η Ουγγρική, η Πολωνική και η Προεδρία της Δανίας και μετά από δύο χρόνια σχεδόν το Συμβούλιο ακόμα δεν έχει θέση επί των προτάσεων του Κοινοβουλίου. Παρ' όλα αυτά, κατά τη διάρκεια της Πολωνικής Προεδρίας είχαμε βάλει και προφορική, συζήτηση, προφορική ερώτηση με συζήτηση στην Ολομέλεια. Στην αρχή της Προεδρίας είχαμε στείλει και μια επιστολή όπου αναφέραμε την προθυμία μας να ξεκινήσουμε ένα άτυπο διάλογο με το Συμβούλιο προκειμένου να βρούμε τις κατάλληλες λύσεις. Καταλαβαίνουμε ότι η κρίση, η οικονομική κρίση δεν ευνοεί τις επενδύσεις σε κοινωνική πολιτική. Πλην όμως, επίσης θέλουμε να πούμε ότι είναι απαράδεκτο να υπάρχουν χρήματα για όλα και ιδιαίτερα για τις τράπεζες, αλλά όχι για τους ανθρώπους. Μας έχουν φτάσει διάφορα μηνύματα για το ζήλο της ε, Κυπριακής ε, Προεδρίας. Άλλωστε, αυτό μας το επιβεβαιώσατε και εσείς σήμερα με τις παρεμβάσεις. Συνεπώς, ε, έχουμε πολλές προσδοκίες από την Κυπριακή Προεδρία. Θα θέλαμε λοιπόν Κομισιόν, Προεδρία και Κοινοβούλιο να κάνουμε ό,τι μπορούμε και θα ήθελα να σα ρωτήσω τι μπορούμε να κάνουμε για να ξεμπλοκάρουμε αυτό το θέμα και το Συμβούλιο να δώσει ένα θετικό μήνυμα. Οι ευρωπαϊκές οικογένειες, οι γυναίκες της Ευρώπης δεν καταλαβαίνουν που το Συμβούλιο δεν λέει τίποτα και παραμένει σιωπηλό για αυτό το θέμα. Καλή επιτυχία στην Προεδρία σας. Eh, σας ευχαριστώ. Και τώρα παρακαλώ τους δύο υπουργούς να λάβουν το λόγο για να μας απαντήσουν. Δυστυχώς δεν έχουμε απεριόριστο χρόνο γιατί έχει προβλεφθεί η ψηφοφορία στις 10.30 ε, ακριβώς, 10 λεπτά. Επομένω θα σας παρακαλέσω να είστε όσο το δυνατόν πιο ε, σύντομοι στις απαντήσεις σας και συνεκτικοί και ίσως ε, μπορείτε να δείτε όλες αυτές τις ερωτήσεις ε, ως ένα δείγμα του πόσο η Επιτροπή μας είναι στρατευμένη στον αγώνα για την ισότητα των δύο φύλων. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο σύντομος μπορώ. Φυσικά πρέπει να δοθούν και οι ανάλογες απαντήσεις, οι διευκρινιστικές. Ε, όσον αφορά η μία ερώτηση και η, πιο εύκολη ερώτηση ήταν πότε θα γίνουν οι σαντήσεις αυτές στην Κύπρο όσον αφορά τα συμφούλια. Η μία θα γίνει, θα λάβει χώρα στις... Ε, ναι. θα γίνει το συνέδριο για τη βία, οικογενειακή βία, θα γίνει στις 8 και 9 Νοεμβρίου του 2011 στη Λευκοσία. Η Λευκοσία είναι η πρωτεύουσα της Κύπρου, όσοι δεν έχετε επισκεφθεί την Κύπρου. Το άλλο συμβούλιο το οποίο, ε, συνέδριο το οποίο θα είναι, θα είναι στη Λευκοσία πάλι 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Και το έναν το οποίο αρμόδιο είναι του Υπουργείου Εργασία και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Θα, θα λάβει η χώρα στη Λεμεσό, μια πολύ όμορφη παραθαλάσσια πόλη, στις 29 και 30 Οκτωβρίου. Όσον αφορά την ερώτηση τι κάνουμε για τη βία κατά των γυναικών. Έχω αναφε... Εκτός τα όσα ε, έχω αναφέρει προηγουμένως, αρχικά πρέπει να πω ότι τα τελευταία χρόνια σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει σημειωθεί πολύ μεγάλη πρόοδο στον τομέα αυτό ως αποτέλεσμα της συνεργασίας του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αναφέρω για παράδειγμα το πρόγραμμα Δάφνη την οδηγία για την εμπορία προσώπων και την οδηγία για το Ευρωπαϊκό Διάταγμα Προστασίας. Επίση, πολύ σημαντική εξέλιξη την οποία χαιρετίζουμε είναι η επίτευξη συμφωνία μεταξύ του Ευρωκοινοβουλίου και του Συμβουλίου σε σχέση με την οδηγία για την προστασία των στην οποία μάλιστα ενσωματώνεται και η διάσταση του φύλου. Παρ' όλα αυτά, οι προσπάθειε και ο αγώνα θα πρέπει να εστιάσουν θα πρέπει να εστιαστούν και όπως ανέφερα και στην ομιλία μου θεωρώ είναι πολύ σημαντικό πέραν των νομοθετικών μέτρων να διαμορφωθεί μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την κατεπολέμηση της βίας ενάντια, εναντίον των γυναικών η οποία θα αποτελεί το γενικό κοινό πλαίσιο πολιτικής για όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαφώτιση για το πρόβλημα της βίας κατά των γυναικών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο είναι πάρα πολύ σημαντική και θα πρέπει να εντατικοποιηθεί, προσφέροντας ταυτόχρονα και τους αναγκαίους πόρους έτσι ώστε να είναι αποτελεσματική. Η καθιέρωση του έτους 2015 ως Ευρωπαϊκού έτους καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών θα συμβάλλει πιστεύουμε καθοριστικά στην ανάδειξη της σοβαρότητας του προβλήματος της βίας και της συστράτευσης που πρέπει να επιτευχθεί για αντιμετώπιση του προβλήματος θα προωθήσουμε τα θέματα αυτά μέσω των συμπερασμάτων του Συμβουλίου. Όσον αφορά το θέμα ε, ποσόστοσης που έχει τεθεί. Σαν Προεδρία υποστηρίζουμε την αυτορύθμιση σαν Κύπρος στον τομέα αυτό και πιστεύουμε ότι μέτρα σε θελοντική βάση μπορεί να προωθηθούν με επιτυχία. Η εισαγωγή ποσοστώσεων παρόλο που έχει αξιολογηθεί θετικά σε ορισμένε χώρε δεν υποστηρίζεται γενικά στην Κύπρο. Η Κύπρο θεωρεί όπω και πολλέ άλλε χώρε μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση ότι το πρόβλημα που υπάρχει μπορεί να επιληθεί όχι μόνο μέσω νομοθετικών μέτρων όπω έχω αναφέρει και προηγουμένω και ρυθμίσεων αλλά στη βάση κατάλληλων μέτρων πολιτική συνοδευόμενων με συγκεκριμένου στόχου. Μερικά παραδείγματα μη νομοθετικών μέτρων που μπορούν να ληφθούν προ την κατεύθυνση αυτή είναι η υιοθέτηση και εφαρμογή συστάσεων σε συγκεκριμένου στόχου σε σχέση με το ποσοστό των γυναικών και των ανδρών στα διοικητικά συμβούλια εταιριών. Η αύξηση της ευαισθητοποίησης των επιχειρήσεων και των εργοδοτών σχετικά με τη σημασία της αύξησης των αριθμών των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις για την ύπαρξη και την, ε, για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα. Και τρίτον, η εισαγωγή κινήτρων για τους κοινωνικούς εταίρους και τις επιχειρήσεις για την εφαρμογή των συγκεκριμένων μέτρων. Όσον αφορά τη σύμβαση προσχώρηση στη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη βία κατά των γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία, Έχουμε δει το θέμα σε Υπουργική Επιτροπή η Υπουργική που ε, ε, έλαβα μέρος ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Υπουργός Εργασίας ε, με όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες οι οποίες ανέλαβαν να μελετήσουν και να αξιολογήσουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση αυτή με βάση την οποία θα ληφθεί και τελική απόφαση η νομοθεσία και οι πολιτικέ μα είναι ευθυγρασμισμένε σε μεγάλο βαθμό με τι πρόνοιε τη Σύμβαση και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια. Ε, να σα πω ότι το βλέπουμε πάρα πολύ θετικά και η Υπουργική Επιτροπή, αφού λάβει υπόψη τη όλε αυτέ τι εκθέσει που ετοιμάζονται και σύντομα θα τι έχουμε, θα αποφασίσουμε θετικά για την προσχώρησή μα στην Σύμβαση του Συμβουλίου τη Ευρώπη. Ε, όσον αφορά το θέμα ε, το θέμα της εμπορίας προσώπων. Η Κυπριακή Προεδρία θα προωθήσει προσχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου ΔΕΗ, το οποίο θα υποβληθεί για ψήφιση στο Συμβούλιο ΔΕΗ τον ερχόμενο Οκτώβριο. Επιπλέον, το συνέδριο που διοργανώνει η Κυπριακή Προεδρία είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε εντάξει στι προτεραιότητε μα αυτό. Για την εμπορία θα αποτελέσει το εφαλτήριο για την υλοποίηση τη νέα στρατηγική κατά τη εμπορία προσώπων, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στι Βρυξέλλε στις 18 Οκτωβρίου του 2012, που είναι η έκτη πανευρωπαϊκή μέρα κατά τη εμπορία προσώπων, όπου θα συμμετέχουν εκπρόσωποι από τα κράτη-μέλη τοπική αλλά και ευρωπαϊκή και διεθνής μη κυβερνητικοί οργανισμοί. Παρούσα στο συνέδριο θα είναι η Υπουργό Εσωτερικών η κυρία Μαύρου και η συντονίστρια τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη εμπορία προσώπων η κυρία Μύρια Βασιλιά. Όσον αφορά, κύριε Πρόεδρε, και τελειώνω νομίζω όσον αφορούν τις, τις, ε, τις μου παρεμβάσεις διευθυνήσεις, ε, όσον αφορά το, τη χρηματοδότηση. Τα χρηματοδοτικά προγράμματα που καλύπτουν θέματα βίας κατά των γυναικών. Όπως έχω ήδη αναφέρει σε ό,τι αφορά την μελλοντική χρηματοδότηση δράσεως στον τομέα της βίας κατά των γυναικών, το Συμβούλιο κατέληξε στις 8 Ιουνίου 2012 σε μερική γενική προσέγγιση επί της σχετικής πρότασης κανονισμού. Το κείμενο περιλαμβάνεται, κείμενο περιλαμβάνεται σαφώς και η χρηματοδότηση δράσεων που να καλύπτουν και θέματα της ε, διάστασης των δύο φύλων αλλά και της προστασίας των θυμάτων. Συγκεκριμένα η πρόταση κανονισμού με βάση την οποία θα επιδιωχθεί συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση με το Ευρωκοινοβούλιο μέχρι το τέλος του χρόνου διαλαμβάνει τα ακόλουθα. Το θέμα της απόδοσης μεγαλύτερης έμφασης στη διάσταση της ισότητας των φύλων και της απαγόρευσης των διακρίσεων. Επισημαίνεται ότι ο τίτλος του προγράμματος έχει αναδιατυπωθεί και περιλαμβάνει τώρα και τη λέξη ισότητα. Οι αντικειμενικοί στόχοι έχουν αναδιατυπωθεί και διασαφινιστεί για να περιλαμβάνουν και τη διάσταση της ισότητας των φύλων, την πρόληψη του ρατσισμού, τη ξενοφοβίας και άλλων μορφών μυσαλλοδοξίας την πρόληψη της βίας κατά των παιδιών, των νεαρών ατόμων και των γυναικών, καθώς και την προστασία θυμάτων και ομάδων κινδύνου. Η πρόταση διατηρεί την αρχή ότι η χρηματοδότηση θα πρέπει να είναι δυνατή για όλους τους πιθανούς δικαιούχους χωρίς διακρίσεις και σε ισότιμη βάση. Όπως έχω ήδη αναφέρει στην, ε, παρουσίαση μου, η Κυπριακή Προεδρία θα συνεχίσει να προωθεί τη διασφάλιση της διάστασης του φύλου και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο σημαντικό ζήτημα των υπηρεσιών στήριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας. Επιπρόσθετα τονίζεται ότι στο πλαίσιο των συμπερασμάτων του Συμβουλίου που θα προωθήσουμε για τη βία κατά των γυναικών, τα οποία στοχεύουμε όπως υιοθετηθούν από το Συμβούλιο Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υποθέσεων, τον ευχόμενο Δεκέμβρη, θα προωθηθεί ξανά η ανάγκη για διασφάλιση επαρκών ευρωπαϊκών πόρων για την ισότητα ανδρών και γυναικών και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών στα πλαίσια του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020. Νομίζω τελειώσαμε. Νομίζω έχω τελειώσει κύριε Πρόεδρε όσον αφορά το δικό μου μέρος. Ναι. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει φοβερή πίεση χρόνου, γι' αυτό θα προσπαθήσω να ομαδοποιήσω ε, τις ερωτήσεις. Ε, το πρώτο που θα ήθελα έτσι να υπογραμμίσω είναι ότι μέσα σε αυτές τις δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες, όπου όλες οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγκαζόμαστε να δούμε και να ξαναδούμε τους προϋπολογισμούς μας για να υπάρξει δημοσιονομική πειθαρχία, είναι ιδιαίτερα σημαντικό η κατανομή των πόρων να γίνει με τέτοιο τρόπο έτσι που να συνεχίσουν να στηρίζονται τόσο μέσα από τους εθνικούς προϋπολογισμούς, αλλά και με την αξιοποίηση των πόρων που η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει στην κατεύθυνση της στήριξης των πολιτικών απασχόλησης προς τις γυναίκες και των πολιτικών κοινωνικής προστασίας. Αυτή είναι μια ευθύνη των κρατών μελών, αλλά είναι και συλλογικά ευθύνη όλων μας, ιδιαίτερα κατά τη διαδικασία του πολιε... της διαπραγμάτευσης του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου, να υπάρξουν εκείνοι οι πόροι, τόσο μέσα από το ε, Ευρωπαϊκό Ταμείο, ε, το Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής, αλλά και μέσα από άλλες πολιτικές, που να στηρίξουν την απασχόληση των γυναικών και την επιχειρηματικότητα των γυναικών, γιατί η στήριξη της επιχειρηματικότητας είναι ένας καλός μηχανισμός για την προώθηση και της απασχόλησης και της ισότητας και της ανέλυξης ε, των γυναικών σε θέσεις ε, κλειδιά στον επιχειρηματικό ε, τομέα. Προς αυτήν την κατεύθυνση θα έλεγα ότι η διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και η αναχώραση στάσης. Είναι σωστόν και καλόν και αυτή θα είναι η δική μας η προσπάθεια να αξιοποιηθούν για να περιληφθεί πλήρως η ενσωμάτωση της αρχής της ισότητας. Ακριβώς έχοντας ε, ως προτεραιότητα την ενίσχυση των συμμετοχικών διαδικασιών σε ό,τι αφορά την υλοποίηση της στρατηγικής Ευρώπη 2020 στην εφαρμογή των κοινωνικών στόχων της στρατηγικής, ειδικότερα της αύξησης της απασχόλησης και της καταπολέμησης της ε, φτώχειας. μία από τις προτεραιότητες που έχουμε θέσει στο Συμβούλιο Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής είναι το πώς δραστηριοποιούμε ακόμα περισσότερο τους κοινωνικούς εταίρους, την κοινωνία πολιτικών και τι αρχέ τοπική διαδικασία εφαρμογή τη στρατηγική, αλλά και στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Και προ αυτή την κατεύθυνση θα έχουμε ειδικό εργαστήριο στο Αντιποσυμβούλιο Συμβούλιο Υπουργών Απασχόληση για να συζητήσουμε αυτό το ειδικό θέμα. Πιστεύουμε ότι μέσα από τι εμπειρίε των δύο τελευταίων χρονιών με την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου μπορούμε να εξάξουμε τα ανάλογα συμπεράσματα έτσι που αυτή η διαδικασία να είναι και όσο το δυνατό πιο συμμετοχική και πιο αποτελεσματική προς την κατεύθυνση της υλοποίηση των στόχων μας για την αύξηση της απασχόλησης και την καταπολέμηση της φτώχειας. Σε ό,τι αφορά το ερώτημα για την ε, φτώχεια για τα παιδιά, ε, προγραμματίζουμε την έκδοση συμπερασμάτων Συμβουλίου για το θέμα της ε, καταπολέμησης της φτώχειας ανάμεσα στα παιδιά και γενικά για το θέμα της ευζοίας ανάμεσα στα παιδιά. Θα χτίσουμε πάνω στη δουλειά ε, που έχει γίνει από μια υπεπιτροπή της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας και αναμφίβολα όλο, αν θέλετε, το έργο που έχει παραχθεί, είτε για επιμέρους πτυχές, είτε συνολικά για αυτό το θέμα, θα αξιοποιηθεί διότι ε, πραγματικά πιστεύουμε ότι είναι ένας τομέας στον οποίο χρειάζεται να δώσουμε ε, μεγαλύτερη ε, έμφαση. Σε ό,τι αφορά διαφορά, τα θέματα της ισότητας της αμοιβή, θα συμφωνήσω απόλυτα ότι μέσα από μια συλλογική προσπάθεια έχουμε παράξει ένα πολύ αξιόλογο νομοθετικό πλαίσιο σε ό,τι αφορά τα θέματα της ισότητας και είναι ταυτόχρονα εξίσου σημαντικό, αξιοποιώντας και τον, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Δύο Φύλων, να εφαρμόσουμε διαδικασίες αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας αυτού του νομοθετικού πλαισίου. Ε, ένας, αυτός θα είναι και ένας επιμέρους στόχος στόχους του τριμερούς συνεδρίου που θα πραγματοποιήσουμε, δηλαδή με τη συμμετοχή των κυβερνήσεων, των εργοδοτικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων στην Κύπρο, όπου θα υπάρξει και ειδική σύνοδος που θα αναφέρεται στο νομοθετικό πλαίσιο, στους μηχανισμούς εφαρμογής και την ε, αποτελεσματικότητά του. Ταυτόχρονα μέσα από το συνέδριο θέλουμε να αναδείξουμε και μέσα από τις εθνικές πρακτικές εκείνες τις θετικές εμπειρίες που μπορούν να βοηθήσουν χώρες μέσα από αυτήν την ανταλλαγή πρακτικών ε, να προχωρήσουν πιο μπροστά σε αυτό το εξαιρετικά ευαίσθητο κεφάλαιο για το θέμα της, ε, της ισότητας. Και θα κλείσω με το θέμα της μητρότητας. Αναφίβολα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο φάι και γίνεται ακόμα πιο δύσκολο σε περιόδους οικονομικής ε, κρίσης. Ε, εκείνο το οποίο θέλω απλά να υπογραμμίσω είναι ότι ξεκινώντας από τη βασική αρχή ότι χρειάζεται να δώσουμε ένα αποτελεσματικό πλαίσιο προστασίας στις έγκυες γυναίκες. Κατανοώντας το γεγονός ότι και στο επίπεδο του Συμβουλίου υπάρχουν μεταξύ των κρατών μελών διαφορετικές προσεγγίσεις γύρω από αυτό το θέμα, νομίζω ότι και έχουμε όλη την καλή διάθεση να επικεντρωθούμε στο κύριο. Και το κύριο είναι να προχωρήσουμε ένα βήμα μπροστά από αυτό στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα, καταλαμβάνοντας υπόψη και τις ευαισθησίες που υπάρχουν σε κράτη-μέλη για αυτό το θέμα, αλλά και το πώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τοποθετείται γύρω από το θέμα της μητρότητας. Θα ήθελα απλώς να κλείσω με μια προσωπική δέσμευση. Η προσωπική μου η δέσμευση είναι ότι θα φροντίσω ε, σε προσωπικό επίπεδο, με, προσωπι... με διμερείς επαφές, να συζητήσουμε κατηδίαν αυτό το θέμα, τόσο με το Ευρωκοινοβούλιο αλλά και με συναδέρφους μου στο Συμβούλιο, για να διερευνήσουμε τις δυνατότητες να ξεκινήσουμε και να προχωρήσουμε σε αυτό το ευαίσθητο και δύσκολο κεφάλαιο. Ευχαριστώ πολύ. Eh, σας ευχαριστούμε, σας ευχαριστούμε πραγματικά πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Λουκά, κύριε Χαραλάμπου. Σας ευχαριστούμε πολύ που αφιερώσετε όλο αυτό το χρόνο στην Επιτροπή μας. Λυπάμαι πραγματικά που δεν είχαμε την δυνατότητα να έχετε το χρόνο να απαντήσετε όλες τις ερωτήσεις. Ξέρετε ότι πρέπει να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία μα. Ψηφοφορίες γίνονται επίση σε πάρα πολλέ κοινοβουλευτικέ επιτροπέ, επομένω πιέζει πολύ ο χρόνο. Όπως είδατε υπάρχουν ορισμένα μέλη της Επιτροπής μας, πρέπει να πάνε και σε άλλε επιτροπέ. Για άλλη μια φορά σα ευχαριστώ ολόθερμα για την παρουσία σα εδώ σήμερα. Πραγματικά προσβλέπουμε σε μια θετική στενή συνεργασία με εσά και βέβαια θα κάνουμε κάθε τι το δυνατό προκειμένου να σα ευχαριστήσουμε, να σα υποστηρίξουμε, συγχωρείτε, στην εργασία που κάνετε για την ισότητα των φίλων. Σας ευχαριστώ και πάλι πολύ. Ας περάσουμε στο σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Συγγνώμη για την καθυστέρηση. Θα καταφέρουμε φαντάζομαι να καλύψουμε τον χρόνο που έχουμε χάσει. Πρωτού ξεκινήσουμε όμως με τις ψηφοφορίες, θα ήθελα να σας ανακοινώσω με ιδιαίτερη ευχαρίστηση ότι ο συντονιστής του ΕΛΚ, η συντονίστρια του ΕΛΚ παντρεύτηκε πρόσφατα. Χαίρομαι πάρα πολύ για σας. Συγχαρητήρια. Σας εύχομαι δύο ανθόσπαρτο. Χαίρομαι πάρα πολύ για σας Από διοικητικής πλευράς όμως ενδεχομένω να υπάρχει πρόβλημα γιατί έχει αλλάξει επίθετο. Κυρία Γκαμπριέλ πρέπει να σας αποκαλώ πλέον και όλοι πρέπει να σας αποκαλούμε κυρία Γκαμπριέλ. Και πάλι συγχαρητήρια. I also just out that Mrs. been married. Και η κυρία Κλέμος επίσης παντρεύτηκε πρόσφατα καταπληκτικά. Συγχαρητήρια και σε εσά λοιπόν. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τις ψηφοφορίες. Πάμε στην πρώτη ψηφοφορία. Κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γερόκα Νέντελζεβα. Πέντε τροπολογίες έχουμε. Μπορούμε να τις ψηφίσουμε από κοινού. Ομπλόκ. Πολύ ωραία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Στην κυρία Γιάροκα μας θα δώσω αυτή τη στιγμή την Προεδρία. Με ιδιαίτερη χαρά μπορούμε να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία για την έκθεσή σας κύριε Γκούσταυσον, ο ρόλος των γυναικών στην φιλοπεριβαλλοντική οικονομία. Θέλετε το λόγο κύριε Πρόεδρε. Ναι, ναι, πολύ σύντομα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετείχαν στην όλη διαδικασία από τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις, από το κοινό. Να ευχαριστήσω βέβαια τους κοιόδης ηγητές και όλο το προσωπικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία σας. Η έκθεση αυτή βελτιώθηκε πάρα πολύ με τις δικές σας τις προτάσεις και να ευχαριστήσω όλος ιδιαιτέρως την Ασάντα και τη Μάλινα, τους βοηθούς μου και τον Σάλταν, ο οποίος με βοήθησε πάρα πολύ στη σύνταξη των συμβαστικών τροπολογιών. Σας ευχαριστώ πολύ για τη βοήθειά σας. Πολύ ωραία. Παράγραφος 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος, παρακαλώ. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 15 για την παράγραφο 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 19 υπέρ. Κατά. Απο... Εγκρίνεται. Αποχές, με συγχωρείτε. Εγκρίνεται. Τροπολογία 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 21. Για την παράγραφο 5β. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Περνάμε στη συμβαστική τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 23. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασική τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 28 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος, άρτη ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Καταπίπτει μάλλον, με συγχωρείτε. Τροπολογή 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 33 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 34 υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονικός έλεγχος για τροπολογία 34, πρόκειται για διαγραφή, άρτη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 39 υπέρ. Κατά αποχές εκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ, κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την ε, συμβαστική τροπολογία 5, άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 13 υπέρ, 10 κατά. Περνάμε στην τροπολογία 43 υπέρ. Κατά. Αποχές Υπέρ για την τροπολογία 43 παρακαλώ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρτε ψηφοφορία για την τροπολογία 43. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 53 υπέρ. Κατά. Στον κατάλογο ψηφοφορίες ε, υπάρχει προφορική τροπολογία. Δεν υπάρχει αντίρρηση. Μπορούμε να ψηφίσουμε. Δεν υπάρχει αντίρρηση. Ψηφίζουμε υπέρ της 53 κατά. Αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ. Το πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της 54 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Παράγραφος 23. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 55. Πρόκειται για διαγραφή υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 8. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 58. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 60 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 60 άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 61 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 61. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Δεν έχει ψηφίσει ένα άτομο, νομίζω Ας επαναλάβουμε την ηλεκτρονική ψηφοφορία, παρακαλώ πολύ, για την τροπολογία 61, άρτη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 9, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβασική τροπολογία 10 υπέρ. Κατά. απόχέ, εγκρίνεται. Τροπολογία 66 υπέρ. Κατά. αποχέ, εγκρίνεται. 67 υπέρ. Κατά. Αποχέ, εγκρίνεται. 68 υπέρ. Κατά. Αποχέ, εγκρίνεται. 69 υπέρ. Κατά. αποχέ, εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. αποχέ, εγκρίνεται. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8 κατά καταπίπτει. Τροπολογία 9 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 10 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 11 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία για την έκθεση αυτή ηλεκτρονική ψηφοφορία. παρακαλώ πολύ, χρησιμοποιήστε τις κάρτες σας, άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με πλειοψηφία. Συγχαρητήρια στον εισηγητή μας. Σας ευχαριστώ πολύ. ευχαριστώ πολύ που αναλάβατε να προεδρεύσω στο κομμάτι. Και τώρα πάμε στην επόμενη ψηφοφορία για τις συνθήκες εργασίας των γυναικών στον τομέα των υπηρεσιών. Ε, ρωτώ πρώτα την εισηγήτρια αν θέλει να λάβει το λόγο, κυρία Γκαρσία Πέρες. Ναι, θα ήθελα να επαναλάβω τις ευχαριστίες σε όλους τους αδέλφους μου που με τις ε, τροπολογίες τους βελτίωσαν την έκθεση αυτή. Είναι μια σημαντική έκθεση. Σχετίζεται με πολύ θεμελιώδη θέματα σχετικά με την ισότητα των γυναικών στην αγορά εργασίας και την συμμετοχή της σε κλάδους και τομείς που η συμμετοχή της είναι πολύ σημαντική. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τους κοιότητες για τη συνεργασία τους και την ε, γραμματεία της ε, Επιτροπής, ε, καθώς επίσης και την βοηθό μου. Καθώς. Αρχίζουμε την ψηφοφορία λοιπόν. Τροπολογία 29 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τώρα πάμε στην 33 υπέρ, κατά, άποχες. Ας επαληθεύσουμε τη 33 παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεν ψηφίζουμε την ε, παρατήρηση για το 2β της απασχόλησης, γιατί αντισωματώνεται χωρίς προφορία. Στη συμβαστική 11 παρακαλώ υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. 36 υπέρ κατά. Αποχές. Ας επαληθεύσουμε την 37 λέει ο πρόεδρος. Πέρας. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται. 67 καταπίπτουν, 39 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 40 σε τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η έξι της απασχόλησης. Το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ας την επαληθεύσουμε. Άρχεται η Εγκρίνεται. 13 συμβαστική υπέρ. Κατά. αποχές εγκρίνεται. Και άρα καταπίπτουν ε, πολλές τροπολογίες και περνάμε στην 14 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Επαληθεύουμε την 52. Επαληθεύουμε την 52 παρακαλώ, άρχεται ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Στη 15, συμβαστική 15 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 4 της Επιτροπής Απασχόλησης ε, δεν ψηφίζεται. 16 τώρα, συμβαστική 16 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 62 υπέρ κατά αποχές. Νομίζω ότι πρέπει να επαληθεύσουμε την 62. Άρχεται η ψηφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. 64 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11, 12, 13 τις απασχόλησης που συμπεριλαμβάνονται χωρίς ψηφοφορία και έτσι πάμε στη συμβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 70 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 71 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 7 της επασχόλησης υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 72 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 73 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, Συμβαστική 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 26 συμβαστική 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 και 3 της Επιτροπής Απασχόλης χωρίς ψηφοφορία ενσωματώνονται και πάμε στη συμβαστική 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 81 υπέρ κατά αποχές. Πρέπει να επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Και πάμε στην 21 συμβαστική υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 15 της απασχόλησης προφορία. Πάμε στη συμβαστική 22 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. ...89 υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται, 90 υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται, 23 συμβαστική υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. Τέσσερα απασχόλησης χωρί προφορία. Συμβαστική 24 παρακαλώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 99 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Α επαληθεύσουμε την 99. Άρχεται η ψηφοφορία. 99. Εψήφισαν όλοι. Όχι ακόμα σας. Είχαμε έναν περισσευούμενο, πρέπει να ξαναγίνει η ψηφοφορία. Άρχεται και πάλι η ψηφοφορία για την τροπολογία 99. Πέρασε. Απερίφθη. Τώρα πάμε στην ε, υπαριθμόν 100 παρακαλώ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 101 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Απασχόληση 9 συμπεριλαμβάνεται χωρίς ψηφοφορία. Πάμε στην τροπολογία 102 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 17 της απασχόλησης που συμπεριλαμβάνεται χωρίς, τροπολο... χωρίς ψηφοφορία. Συμβαστική υπαριθμών 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται β και γ, β και σ εσυμματώνονται είναι της απασχόλησης. Πάμε συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά άποχες. Εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 9 παρακαλώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική παριθμών 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8, συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ κατά αποχές Πρέπει να επαληθεύσουμε νομίζω για την 24 άρχεται η ψηφοφορία. 24 πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Υπάρχει μόνο ένα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δύο υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται και τώρα όλο το ψήφισμα με ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχιτη ψηφοφορία. Είναι προφανές ότι υιοθετήθηκε και επομένως ευχαριστούμε και συγχαρητήρια στην κυρία Συγήτρια. Θα συνεχίσουμε σε ένα λεπτό. Παρακαλώ καθίστε. Ίσως ξέχασα να σας το πω. θα σας το υπενθυμίσω ότι το σημείο 8 αναβλήθηκε για τις 3 Σεπτεμβρίου. Οπότε θα περάσουμε κατευθείαν στο 9. Οπότε γυρίζω ξανά στα Σουηδικά. Έχει λήξει η ψηφοφορία. Περνάμε στο σημείο 10 της διάταξης. Συγγνώμη, 9 λέει ο πρόεδρος. Εξάλληψη των συνδεόμενων με το φύλλο στερεοτύπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτο προσχέδιο από την κυρία Λιωτάρ. Έχετε το λόγο. Ja, dank u wel, voorzitter. En als u in het Ε, μετά τα δικά σας ε, σουηδικά πρόεδρε θα μιλήσω και εγώ ολλανδικά λοιπόν. Αφού όλοι φορούν τα ακουστικά ήδη. Θα ακολουθήσω το δρόμο σας. Χαίρομαι που είναι παρούσες και παρόντες το συνάλφοι. Χρειάζομαι τη βοήθειά σας για να βελτιώσω το κείμενο στην κοινωνία μας. Σε πολλούς τομείς και σε πολλά επίπεδα εξακολουθούν να υφίστανται στερεότυπα σχετικά με το φύλλο το, ε, και την θέση των γυναικών και των ανδρών. Είναι τόσο συχνά αυτά τα στερεότυπα που μα, πολλές φορές διαφεύγουν της προσοχής μας. Όμως τα στερεότυπα ε, επηρεάζουν ε, σε μεγάλο βαθμό τις ευκαιρίες που μας δίδονται και το μέλλον μας, όλων, ανδρών και γυναικών. Ιδιαίτερα όμως για τις ε, γυναίκες οι επιπτώσεις αυτής της κατάστασης είναι πολύ πιο βαριές και αρνητικές από ότι η επιπτώση των ανδρών. Η ύπαρξη στερεοτύπων ε, είναι, βρίσκεται παντού στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στον τύπο, την τηλεόραση, τις διαφημίσεις και στην εκπαίδευση πολλές φορές, στα βιβλία. Έχουμε βιβλία μαθημάτων που παρουσιάζουν τους άντρες και τις γυναίκες με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Μετά, οι κοινωνίες επίσης ε, προσδοκούν από τις γυναίκες να αναλάβουν συγκεκριμένους ρόλους, για παράδειγμα της νοικοκυράς, ε, ή της μητέρας. Αυτό προφανώς όλα αυτά επηρεάζουν τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας που έχουν οι γυναίκες. Και για τους άνδρες και αυτό, διότι και οι άνδρες πολύ συχνά ε, είναι υποχρεωμένοι σε εισαγωγικά να εργάζονται σε συγκεκριμένα επαγγέλματα ε, και όχι σε επαγγελμάτα που θεωρούνται γυναικεία. Το 2011 στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση οι γυναίκες επίσης ε, ε, κερδίζουν 16,4% λιγότερο από ότι άντρες για την ίδια δουλειά. Η παρουσία τους είναι, πολύ, είναι μικρότερη και σε διευθυντικές θέσεις επιχειρήσεις και στον δημόσιο τομέα αν φανταστούμε ότι, αν λάβουμε υπόψη ότι οι γυναίκες εκτός από τη δουλειά κάνουν και έχουν και άλλες υποχρεώσεις, οικογενειακές και άλλες, ε, εργάζονται σε μεγαλύτερο, καταλαβαίνουμε γιατί εργάζονται σε μεγαλύτερο βαθμό, ε, σε πιο ε, προσωρινές θέσεις εργασίας, με ένα ωράρια κλπ. Αυτό της ε, οδηγεί σε μεγαλύτερο κίνδυνο να περάσουν στη φτώχεια τη στιγμή της σύνταξης. Συντάξεις τώρα. Η διαφορά των συντάξεων ανάμεσα σε γυναίκες και άντρες είναι γνωστή. Οι γυναίκες επιβαρύνονται μάλιστα από την Λευκή Βίβλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλώ για τη Λευκή Βίβλο στην έκθεσή μου. Πιστεύω ότι χρειάζεται καινούρια νομοθεσία που θα επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτά τα στερεότυπα και τις ανισότητες ανάμεσα στις γυναίκες και τους άντρες. Νομοθεσία η οποία θα καταπολεμήσει τα στερεότυπα που είναι τόσο πολύ επίμονα στις κοινωνίες μας. Η έκθεσή μου περιορίστηκε σε τέσσερις σελίδες, παρόλο που θα ήθελα να είναι περισσότερες. Αναφέρω σε ποιους τομείς υπάρχουν πολλά στερεότυπα, μέσα ενημέρωσης, διαφημίσεις, ε, εργασίας, λήψη πολιτικών αποφάσεων. Μίλησα για, τις, ε, για τη δράση Ευρωπαϊκής, ε, μίλησα για τη λήψη οικονομικών και πολιτικών αποφάσεων, για τη δράση Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάνω κάποιες προτάσεις στους νομοθέτες στον νομοθέτη για να βελτιωθεί η κατάσταση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν μπαίνω σε πάρα πολλές λεπτομέρειες στην έκθεσή μου. Προσπαθώ να υποβάλω ένα γενικό πλαίσιο και περιμένω από την Κομισιόν να το συμπληρώσει. Περιμένω τις ε, τοποθετήσεις σας για αυτό που γέννησα εγώ στο χαρτί για το πνευματικό μου τέκνο. Θέλω να μου πείτε αν σας αρέσει, αν πρέπει να αλλάξουμε κάποια πράγματα κλπ. Eh, Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Κυρία Λεωτά, είναι ένα θέμα ιδιαίτερα σημαντικό. Ε, τα στερεότυπα επηρεάζουν πάρα πολλά πράγματα στη ζωή των γυναικών. Θα δώσω το λόγο καταρχήν τον κύριο Ταραμπέλα. Θα ήθελα να ε, καθησυχάσω την εισηγητρία, είναι εξαιρετική η έκθεσή της. Ε, αναφέρεται στα στερεότυπα και στην εισαγωγική έκθεση ε, στην αιτιολογική εκθέση και στο διατακτικό. Ε, τα στερεότυπα ε, σε μεγάλο βαθμό οφείλονται στι διαφημίσει και στα μέσα ενημέρωση. Ξεκινάνε από πολύ νωρί στη ζωή των ανθρώπων, τα, από την παιδική ηλικία και είναι πολύ επίμονα. Χαρακτηρίζουν τη συμπεριφορά των ανθρώπων και όταν μεγαλώνουν. Προφανώς τα στερεότυπα τονίζονται και από το σχολείο και από το πανεπιστήμιο και πολλές φορές και στην αγορά εργασίας γιατί ορισμένα επαγγέλματα είναι δεσμευμένα ε, για τους άντρες ή για τις γυναίκες. Ε, για την έκθεση Λιωτά θέλω να πω ότι κατά την άποψή μου είναι περιττό να νομοθετήσουμε. Ήμουν ε, υπουργό ε, στη γαλλόφωνη περιοχή του Βελγίου για μερικά χρόνια και είχαμε σκεφτεί να νομοθετήσουμε και κάθε φορά σταματούσαμε ε, λέγοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση νομοθετεί για αυτά τα θέματα, τότε πρέπει να περιμένουμε να εφαρμόσουμε την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά εμείς. Ε, περάσαμε έτσι πολλά χρόνια διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σταματούσε να νομοθετεί. Ίσως λοιπόν θα διαφωνούσα με την παράγραφο 16 να ενθαρρύνει το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων και τα διάφορα εθνικά ιδρύματα να προωθήσουν την περαιτέρω έρευνα σχετικά με τα βασικά αίτια των στερεοτύπων. Ε, δεν ξέρω αν θα πρέπει να γίνει μια τέτοιου είδου έρευνα. Το σημαντικό είναι να γίνουν ε, εκστρατείε ενημέρωση, ιδιαίτερα στα σχολεία, ε, να γίνει μια ενημέρωση για την ποικιλία των διαφόρων σταδιοδρομιών και επαγγελμάτων που υπάρχουν ε, και αυτό δεν έχει σχέση μόνο με τα στερεότυπα. Ίσως δεν, δίνουν, δεν δίνουμε ε, στα γυμνάσια και στα λύκεια, στα παιδιά επαρκή ενημέρωση για την γάμα των επαγγελμάτων που υπάρχουν ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ε, επιστημονική έρευνα και αυτά τα παιδιά τελειώνουν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και δεν ξέρουν τι να κάνουν στο πανεπιστήμιο γιατί δεν έχουν λάβει επαρκείς πληροφορίες επαγγελματικού προσανατολισμού. Συνεπώ περισσότερες πληροφορίε και καλύτερες πληροφορίε και δράση κατά πολέμηση των στερεοτύπων αντί για έρευνα. Για παράδειγμα, ένα επάγγελμα, ε, οι ηλεκτρόλοι μηχανολόγοι, ε, τεχνικοί, τεχνίτες, που θεωρείται ανδρικό επάγγελμα και άλλα επαγγελματά υπάρχουν τέτοια επαγγελμάτα που οι γυναίκες δεν γίνονται δεκτές. Ίσως θα πρέπει να επιμείνουμε στην ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση, αντί στην έρευνα για τα στερεότυπα. Τα στερεότυπα είναι πολιτιστικά, έχουν ιστορικό υπόβαθρο, οφείλονται και στις ε, σωματικές μας διαφορές. Είμαστε ίσοι ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, αλλά δεν είμαστε ίδιοι όμοιοι. Λοιπόν, περισσότερες δράσεις, ευαισθητοποίησεις, καταπολέμηση των στερεοτύπων, από πιο νωρί. και η κυρία Λεωτάρη έχει δίκιο σε αυτό, ε, επίσης δράση μέσω των μέσων ενημέρωσης, της διαφήμισης του τύπου. Και επίσης και πιο και μεταγενέστερα στη ζωή των ε, νέων όταν ήδη διαλέγουν ένα επάγγελμα στο πλαίσιο της, ε, του χώρου εργασίας. Αυτά, ε, ελάχιστες οι τροπολογίες που θα ήθελα να γίνουν. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ζητώ συγγνώμη, θα δείξω αγένεια πρόεδρε, διότι πρέπει να πάω στην πλατεία του Λουξεμβούργου, εδώ από πίσω, για να συναντήσω του παραγωγού γάλακτο που αντιμετωπίζουν δυσκολίε. Θα πρέπει να καταλήψω την αίθουσα. Συγγνώμη. Σα ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Κλειβέτη έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ την κυρία Λιωτάρ για την έκθεσή της, που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική το έχω πει πολλές φορές ε, ότι δεν συζητάμε επαρκώς, δεν αναλύουμε επαρκώς το ζήτημα των στερεοτύπων, το πρόβλημα των στερεοτύπων και θεωρώ ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε και λίγο περισσότερο με το γεγονός ότι η κοινωνία εν γέννη δίνει πολύ μεγάλη σημασία στα στερεότυπα. Και αυτό το λέω σκεφτόμενοι ότι από τη ε, μία πλευρά θεωρούμε ότι υπάρχει ένα κάποιο ταμπού για τα στερεότυπα αυτά, τα αποδεχόμαστε, αποδεχόμαστε τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν τη σκέψη μας και τη δράση μας. Πολλές φορές όταν ασχολούμαστε με το ζήτημα των ανισοτήτων ανδρών και γυναικών να εντοπίσουμε και τα στερεότυπα αυτά τα οποία είναι πάντα παρόντα και πολλές φορές λειτουργούν σαν απόλυτοι κανόνες και απόλυτοι νόμοι. Και από την άλλη βλέπουμε ότι ε, υπάρχουν και στερεότυπα τα οποία αντιμετωπίζονται ως ε, αιτιολόγηση της ύπαρξης ανισότητας μεταξύ των ανδρών και γυναικών λέγοντας ότι ναι υπάρχουν κάποιοι λόγοι παραδοσιακοί πολλές φορές που εξηγούν την ανισότητα μπορεί να υπάρχει ανάμεσα στα δύο φύλλα. Διαβάζοντας λοιπόν την έκθεση αυτή της κυρίας Λιωτάρ βλέπουμε κάποια κάποιες πολύ καλές προτάσεις αντιμετώπισης του προβλήματος αυτού. Θα μπορούσαμε να βρούμε και άλλες λύσεις. Βλέπουμε ουσιαστικά ότι τα στερεότυπα είναι ένας κοινωνικό κοινωνικός εχθρός που ουσιαστικά μας εμποδίζει πολλές φορές να λάβουμε δράση και να καταπολεμήσουμε, να εξαλείψουμε τις ανισότητες κάτι ακόμα πρέπει να κάνουμε και ως προς αυτό μας βοηθάει και η έκθεση, είναι να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις άμεσες επιπτώσεις των στερεοτύπων όσον αφορά την ανισότητα ανδρών και γυναικών. Γιατί ξέρετε ότι προφανώς θα πρέπει να εντοπίσουμε τους απαραίτητους τομείς και τα απαραίτητα μέσα για να εξαλείψουμε την ανισότητα αυτή. Όταν όμως έχουμε κάποια πολύ συγκεκριμένα μέσα, τότε βλέπουμε ότι εξακολουθούμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα όταν δεν βλέπουμε ποιε είναι οι άμεσε επιπτώσει των στερεοτύπων στην ζωή των ανθρώπων. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω την συνάδελφό μα κυρία Λιωτάρ. Όπως μας είπε επίσης, θέλει τη δική μας συνεργασία για την περαιτέρω βελτίωση της έκθεσης αυτής. Πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνουμε κάθε τι το δυνατό, προκειμένου να καταπολεμήσουμε αποτελεσματικά τα στερεότυπα αυτά, τα οποία καθορίσουν πολλές φορές τη ζωή μας και πιστεύω ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στη σωστή τους διάσταση. Να δούμε δηλαδή ότι πρόκειται ουσιαστικά για νοοτροπίες οι οποίες πρέπει να τροποποιηθούν. Αν μη τι άλλο πιστεύω ότι με την τροποποίηση αυτή θα επέλθει και μια τροποποίηση στο καθεστώς ανισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Σας ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Κυρία Τσοσκουβάη, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την έκθεσή της κατά την άποψή μου εντοπίζεται πραγματικά στα βασικά σημεία που πρέπει να δοθεί η μάχη για την εξάλληψη των στερεοτύπων που αφορούν το φύλλο. Σαφώς θα πρέπει να ασχοληθούμε με τα μέσα ενημέρωσης και τη διαφήμιση. Βλέπουμε στον τομέα αυτό την άνθηση των στερεοτύπων αυτών, στερεότυπα τα οποία μπορούν να πειράσουν τα παιδιά σε πολύ νεαρή ηλικία. Είμαι πεπισμένη όμως ότι ε, ο βασικός ρόλος μπορεί να διαδραματιστεί κυρίως μέσω των γονιών. Οι γονείς είναι αυτοί οι οποίοι δίνουν το παράδειγμα στα παιδιά τους. Θα ήθελα συγκεκριμένα τώρα να αφαιρθώ σε κάποιους τομείς, στους οποίους αναφέρεται και η εισηγήτρια. Παράγραφος 6. Εκπαίδευση και μέσα ενημέρωση. Στο σημείο 6 αναφερόμαστε σε κάποια προγράμματα τα οποία προωθούν αρνητικά στερεότυπα στα μέσα ενημέρωσης. Πώς μπορούμε να κάνουμε την καταμέτρηση, την ανάλυση που προτείνεται εδώ πέρα, ποιος θα είναι ο απότερος στόχος, ποιοι είναι οι δείκτες οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν. Θα ήθελα να ζητήσω από την εισηγήτρια να μας πει τι εννοεί ακριβώς το σημείο 6, σημείο 4. Επαγγελματικός προσανατολισμός. Συμφωνώ με την σχετική πρόταση που γίνεται στο σημείο αυτό αλλά δεν πιστεύω ότι τα τακτικά μαθήματα είναι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Επίσης, δεν γνωρίζουμε ποιος θα χρηματοδοτήσει τα προγράμματα αυτά. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα προγράμματα αυτά. Νομίζω ότι θα μπορούσαν να διεξαχθούν κάποιες εκστρατείες σαν αυτή που έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες υπό τον τίτλο «Γυναίκες και έρευνα». Αγορά εργασία. Συμφωνώ ότι στην αγορά εργασία πολύ συχνά οι γυναίκε πρέπει να αντιμετωπίσουν στερεότυπα, τα οποία οδηγούν σε πολύ σημαντικέ ανισότητε. Ω προ τα σημεία όμω F και G πιστεύω ότι θα πρέπει η διατύπωση να είναι λίγο πιο προσεκτική. ιδίω όσον αφορά τι ευέλικτε ώρε εργασίε. Πολλέ φορέ οι γυναίκε που έχουν παιδιά επιθυμούν να έχουν ευέλικτο ωράριο ή, ε, ή μερική απασχόληση, γιατί αυτό του επιτρέπει πολλέ φορέ να φροντίσουν καλύτερα τα παιδιά του. Στο σημείο G. Η πληροφόρηση που μα δίνεται στο σημείο αυτό δεν είναι αντικειμενική κατά την άποψή μου θα ήθελα να γνωρίζω αν υπάρχουν συγκεκριμένα στατιστικά δεδομένα, τα οποία να καταδεικνύουν ότι όντως οι γυναίκες υποβάλλουν συχνά αιτήσει προκειμένου να εργαστούν ως πυροσβέστες, για παράδειγμα. Υπάρχουν στατιστικά δεδομένα για τις αιτήσει γυναικών σε κατεξοχήν αντρικά επαγγέλματα. Ενδεχομένως να γίνονται άντρες πιο δεκτοί να προσλαμβάνονται πιο συχνά άντρε στι θέσει αυτέ, ακριβώ επειδή οι άντρε είναι τελικά αυτοί που κάνουν αίτηση για αυτέ τι θέσει. Νομίζω ότι ε, το βασικό εμπόδιο πολλές φορές για κάποιες τέτοιες θέσεις εργασίας δεν είναι τόσο οι διακρίσεις, ως το γεγονός ότι οι γυναίκες σωματικά μπορεί να μην ανταποκρίνονται στις ε, θέσεις αυτές εργασίας, όσον αφορά δηλαδή την σωματική δύναμη που απαιτείται. Θα ήθελα να αφαιρθώ σε κάτι ακόμα που πιστεύω ότι θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην έκθεση. Τα στερεότυπα που φερούν το φύλλο εντοπίζονται κυρίως στα παιδιά, ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να σας πω ότι η καταπολέμηση των στερεοτύπων που αφορούν το φύλλο θα πρέπει να υποβοηθηθεί από μία οικογενειακή πολιτική που θα επιτρέπει στις γυναίκες να εξορροπούν σωστά την επαγγελματική και την προσωπική του ζωή. Ενδεχομένως να επαναλαμβάνομαι, δεν είμαι σκιώδης εισηγήτρια, πάντως πιστεύω ότι το ζήτημα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να υπάρχει δηλαδή μια οικογενειακή πολιτική κατάλληλη και γνωρίζουμε ότι η οικογενειακή πολιτική πολύ συχνά αποτελεί αρμοδιότητα εθνική. Στο επίπεδο αυτό λοιπόν βλέπουμε ακόμα ότι υπάρχουν πολλά εμπόδια. Αναφερθώ στο σημείο 14 επίση τη έκθεση. Νομίζω ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα πρόβλημα όσον αφορά την αξιολόγηση και την ανάλυση των στερεοτύπων που αφορούν το φύλλο. Η συγγήτρια πολύ σωστά λέει ότι θα πρέπει εδώ πέρα να αναπτύξουμε περισσότερους δείκτες. Η κατάρτιση όμως των δικτών αυτών θα πρέπει να αποτελεί τμήμα της δραστηριότητας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών και να μην αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε κάθε περίπτωση θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την πολύπλοκη αυτή έκθεση. Αναμφίβολα πρέπει να μιλήσουμε περισσότερο για την εξάλληψη των στερεοτύπων που φορούν το φύλλο και ως προς αυτό θα υποβάλω κάποιες τροπολογίες. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Η κυρία Κορνέλης έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την ε, έκθεση αυτή. Είναι πολύ δύσκολο να βρει κανείς κάτι αρνητικό σε αυτή την έκθεση, γιατί είναι θετική στα περισσότερα σημεία της. Όντως το ζήτημα είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο. Ένα ζήτημα ιδιαίτερα δύσκολο, γιατί πολλές φορές ε, είναι δύσκολο να μιλάμε για την εξάλληψη των στερεοτύπων χωρίς να φτάνουμε τα όρια της ελευθερίας της ε, έκφρασης. Δεν είναι πολύ εύκολο επίσης να πείθουμε τους ανθρώπους κάθε φορά να αλλάζουν μόνοι τους νοτροπία ή κειστάσι. Θεωρώ λοιπόν ότι και στάση. Θεωρώ λοιπόν ότι η διαπαιδαγώγηση και η ευαισθητοποίηση αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μέσα τα οποία διαθέτουμε για το σκοπό αυτό. Και πολύ σωστά αναφερόμαστε επίσης και στις διαφημίσεις. Ένα τομέα στον οποίο παρουσιάζονται πάρα πολλά στερεότυπα που φορούν το φύλλο. Υπάρχουν πάρα πολλές διαφημίσεις για απορριπαντικά, για ηλεκτρικές σκούπες κτλ. Και κάθε φορά που υπάρχει ένας άντρας που συμμετέχει σε μια τέτοια διαφήμιση, ουσιαστικά όταν βλέπουμε έναν άντρα ο οποίος συμμετέχει σε μια διαφήμιση ηλεκτρικής σκούπα, τονίστε πάρα πολύ και η απορροφητική δύναμη της α, α, ηλεκτρικής στην περίπτωση αυτή. Επίσης, Υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο χάσμα όσον αφορά την ισότητα των φύλων εξαιτία των στερεοτύπων. Ένα χάσμα πολύ σημαντικότερο από το χάσμα το οποίο παρουσιάζεται στι αμοιβέ, στου μισθού. Ένα σημείο το οποίο θα μπορούσαμε να προσθέσουμε είναι να δούμε και ποιε είναι οι ίδιε οι ανακοινώσει και εκστρατείε που γίνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θυμάμαι ότι πριν από μερικέ εβδομάδε έγινε μια πολύ μεγάλη εκστρατεία για τα κορίτσια και την έρευνα, όπου στην καμπάνια αυτή χρησιμοποιήθηκαν ω σύμβολα κραγιόν και ψηλοτάκουνα παπούτσια. Και ξέρετε ότι η σελίδα της εκστρατείας αυτής μέσα σε δύο μέρες συγκέντρωσε 8.000 αρνητικές απόψεις. Προφανώς δεν έπρεπε να δεξαχθεί κατά αυτόν τον τρόπο να χρησιμοποιηθούν τουλάχιστον αυτά τα σύμβολα. Έπρεπε να ήμασταν πιο προσεκτικοί. Η καταπολέμηση των στερεοτύπων έχει να κάνει με την δυνατότητα δημιουργίας μιας ελευθερίας επιλογής. Υπάρχουν πολλές γυναίκες και πολλοί άντρες που ουσιαστικά αποτελούν θύμα των στερεοτύπων, δεν έχουν ελευθερία επιλογής εξαιτίας της ύπαρξης στερεοτύπων. Σαφώς μπορεί κανείς, να, μια γυναίκα, να έχει μια πλήρη επαγγελματική καριέρα, να εργάζεται πλήρως, χωρίς να είναι κακή μητέρα αναγκαστικά. Εγώ πολλές φορές πηγαίνω και παίρνω τα παιδιά μου την Παρασκευή α, το βράδυ αφού έχω τελειώσει τη δουλειά μου και βλέπω ότι εντυπωσιάζονται πολλές φορές οι γυναίκες προσέχουν τα παιδιά λέγοντας «Α, τελικά είστε εσείς η μητέρα, μάλιστα». Στις κάτω χώρες πάντως υπάρχουν ε, και αλλού πιστεύω πολλές γυναίκες οι οποίες επηρεάζονται από τα αρνητικά στερεότυπα που υφίστανται για τις γυναίκες που απασχολούνται πλήρω. Πολλά πράγματα πρέπει να γίνουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και πιστεύω ότι υπάρχουν κάποια σημεία στα οποία μπορούμε να δυναμώσουμε ακόμα περισσότερο την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ. Eh, Σας ευχαριστώ. Δεν βλέπω να στείλει σε το λόγο. Όχι, ζητώ συγγνώμη, μήπως κάποιος από την Επιτροπή. Παρακαλώ. να σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, που μου δίνετε το λόγο. Θα ήθελα βεβαίω να ευχαριστήσω την ε, Επιτροπή των Γυναικών και την συγκεκριμένη την κυρία Λιωτάχ για την έκθεση αυτή, η οποία πραγματεύεται ένα θεμελιώδες ζήτημα, ένα θεμελιώδες εμπόδιο ως προς την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, η καταπολέμηση δηλαδή των στερεοτύπων ως προς το ρόλο των φίλων που έχουν παγιωθεί μέσα στην καθημερινή ζωή είναι αγώνα μεγάλο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπογραμμίσατε και σε άλλου ότι αποτελεί μεγάλο εμπόδιο στην ισότιμη μεταχείριση. Ε, νοθεύει το έδαφος ισότιμου ανταγωνισμού, τις ε, φιλοδοξίες, τις προσδοκίες και βέβαια την αξιοποίηση των ε, ιδιαίτερων ικανοτήτων, ε, του ταλέντου δηλαδή, είτε του άντρα είτε της γυναίκας. Και έτσι λοιπόν μέσα στρατηγική για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για την περίοδο 2010-2015 έχει εγγραφεί αυτός ο στόχος κατά πολέμηση των στερεοτύπων. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποιες τροπολογίες, που έχει αναλάβει, πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Μάντρων Στερεοτήτων, των οποίων και εσείς υπογραμμίσατε κυρία Λιωτάχ στην εκθεσή σα κάποιες ε, πρωτοβουλίες που θα αναφέρω, που όμως δεν μπορούν να είναι εξαντλητικές, καθώς δεν έχω το χρόνο σήμερα. Στο χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης κυρίως. Θα ήθελα να επισημάνω ότι στο πλαίσιο της υλοποίησης της πλατφόρμας δράσης του Πεκίνου, η προσεχής Προεδρία, η Ιρλανδία δηλαδή, απεφάσισε να εργαστεί με βάση τον, το, το ρόλο των γυναικών, την παρουσία των γυναικών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και έτσι η επερχόμενη αυτή Προεδρία ε, ζήτησε από το Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων να συλλέξει στοιχεία και να επεξεργαστεί δείκτες ως προς την συμμετοχή των γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης και στα 27 κράτη-μέλη, στην την Κροατία, και να συλλέξει πληροφορίες για τους ε, κώδικες, εθελοντικούς δηλαδή κώδικες, δηλαδή ε, συμπεριφοράς που υιοθετεί ενδεχομένω ο τομέας των ΜΜΕ. Για την εκπαίδευση. Στον χώρο της παιδείας λοιπόν επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω ότι στο πλαίσιο του προγράμματος Κομένιους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει την συνεργασία μεταξύ σχολείων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απάλληψη των στερεοτύπων ανάλογα με το φύλλο και για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι το 2009 στο πλαίσιο ενός προγράμματος ανταλλαγών βέλτιστων πρακτικών ως προς την ισότητα ανδρών και γυναικών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οργάνωσε ανταλλαγές ακριβώς για το θέμα των ε, της καταπολέμησης των στερεοτύπων στα σχολεία έτσι ώστε να δώσουμε την ευκαιρία στα γόρια και στα κορίτσια στο σχολείο να ε, προετοιμαστούν για μελλοντικές επιλογές αργότερα στη ζωή τους, ε, να προετοιμαστούν για ε, επιλογές εκπαιδευτικές στην σχολική τους πορεία που ίσως να μην ήταν αυτές που θα υποδείκνυαν τα στερεότυπα. Και επίσης τον Οκτώβριο του 2012 προτείνουμε μια εκδήλωση κατάρτισης για την εκπαίδευση, κατάρτιση των φύλων για την εκπαίδευση, με την Ισπανία, την Πορτογαλία, τις κάτω χώρες που θα παρουσιάσουν δραστηριότητες που έχουν αναπτύξει, ευαισθητοποίησης δηλαδή των εκπαιδευτικών και των μαθητών για το ρόλο των φύλων για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Και έτσι τα λοιπά και συμμετέχοντα κράτη θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν το ενδεχόμενο να μεταφέρουν αυτές τις εμπειρίες και τις πρακτικές της χώρας τους. Επίσης, το χώρο εργασίας που είναι πολύ σημαντικό στοιχείο, είναι δηλαδή ο χώρος εκείνος στον οποίο ε, πολλαπλασιάζονται τα στερεότυπα για το ρόλο των φύλων. Ε, όπως είπατε και εσείς κύριε Λιωτάρ, δραστηριότητες ευαισθητοποίησης έχουν πολύ μεγάλη σημασία και ιδιαίτερα για να μιλήσουμε για αίτια και κινδύνους της απόκλησης της αμοιβέ μεταξύ ανδρών και γυναικών. Θα σας θυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ηγηθεί μιας εκστρατείας ενημέρωσης ευρείας κλίμακος για την καταπολέμηση των αποκλήσεων μεταξύ ανδρών και γυναικών ως προς αμοιβές του στην περίοδο 2009 με 2012. Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω ότι εφέτος οργανίσαμε τη δεύτερη Ευρωπαϊκή ημερίδα για την καταπολέμηση της, των αποκλήσεων στις αμοιβέ, στους μισθούς, το Μάρτιο εφέτος και βέβαια κάθε χρόνο επιλέγουμε την ε, ημέρα που φέρει τον αριθμό ε, τον αντίστοιχο με αυτόν της μισθολογικής απόκλησης. Δηλαδή πόσες μέρες περισσότερες θα έπρεπε να δουλεύει μια γυναίκα το μήνα για να έχει ισοδύναμο μισθό με αυτό, ε, τον ίδιο μισθό με αυτό του άντρα. Αυτή είναι η μέρα ε, κατά την οποία επιλέγουμε να διεξαχθεί αυτή η μερίδα. Επίσης προχωρούμε και σε μελέτες των αιτίων και των συνεπειών των της απόκλησης αυτής, της μισθολογικής, ενθαρρύνοντας και τις επιχειρήσεις να επιληφθούν του θέματος αυτού. Έχουμε δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και κατάρτισης στο θέμα αυτό. Και ένας από τους σημαντικούς τομείς αν προκειμένου είναι να ενθαρρύνονται οι επιχειρήσεις στην αξιοποίηση του δυναμικού και των ταλάντων των γυναικών στους τομείς εκείνους όπου είναι υπό εκπροσωπούμενοι οι άνδρες. Επίσης, ε, ή μάλλον που είναι εκπροσωπούμενες οι γυναίκες, δηλαδή τομείς αποκλειστικά των ανδρών. Επίση, ε, στον τομέα τη ευαισθητοποίηση, θα γνωρίζετε ασφαλώ ότι το Μάρτιο του 2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προ... Ε, κατέθεσε σχέδιο εκθέσεως για την πρόοδο στο θέμα της συμμετοχής των γυναικών στη λήψη οικονομικών αποφάσεων και δεδομένου ότι κρίθηκαν ανεπαρκείς οι πρόοδοι, αναζητούμε αυτή τη στιγμή διαφορετικές νέες επιλογές, εναλλακτικές επιλογές για μέτρα εστιασμένα στον τομέα αυτών να φτάσουμε σε μια πιο ισορροπή εκπροσώπηση των γυναικών και των δρόμων στη διαδικασία λήψη αποφάσεων, δεδομένου ότι και αυτή είναι μία από τις συνέπειες, αυτό το χαρακτηριστικό είναι μία, μία από τις συνέπειες των στερεοτύπων Ω προ το ρόλο μπορεί να λαμβάνει ένας άντρα ή μια γυναίκα σε μια επιχείρηση σε ένα χώρο εργασία. Θα ήθελα επίση να υπογραμμίσω τρία ζητήματα στο ευρωπαϊκό κοινωνικό μέτωπο που επίσης υπογραμμίσατε ως πολύ σημαντικό στην περίοδο την προγραμματική που τρέχει αυτή την εποχή έχει γίνει μια αξιολόγηση για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τις δράσεις δηλαδή τις οποίες αναπτύξαμε, οι οποίες αναπτύχθηκαν για να αντιμετωπιστούν ε, τα πολιτιστικά και κοινωνικά στερεότυπα. Μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης στη σχετική μελέτη, αν το επιθυμείτε. Η δε προσεχής προγραμματική περίοδος προβλέπεται επίσης να περιλάβει το θέμα αυτό κατά προτεραιότητα. Ε, τις πληροφορίες, όπως είπα, μπορείτε να τις αναζητήσετε στο Staff Working Document, στοιχεία για ένα στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020, έγγραφο το οποίο θετήθηκε από την Επιτροπή το Μάρτιο του 2012. Ο δε ρόλος των, γυναικών, ανδρών τώρα, προτελευταίο σημείο, ο ρόλος των ανδρών Είναι βέβαια ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Ένα από τα οριζόντια θέματα στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική και θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι το 2010 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ξεκίνησε μία μελέτη για το ρόλο των ανδρών προκειμένου να επιτευχθεί στο στόχο της επίτευξης της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Μία μελέτη η οποία θα παρουσιαστεί σε μία διάσκεψη το Σεπτέμβριο του 2012 στις Βρυξέλλες και η οποία ελπίζουμε θα επιτρέψει να ε, παρουσιαστούν προς τρεις πληροφορίες ε, στους αρμόδιους για τη λήψη των αποφάσεων, έτσι ώστε να λαμβάνουν αποφάσεις πιο πολύ για την πρόθεση της δυνατότητας συμμετοχής των γυναικών ε, στην κοινωνία. Υπογραμμίστηκε λοιπόν ο ρόλος της εκθέσεως. Θα ήθελα απλώ να υπογραμμίσω για την Επιτροπή σας ότι το τωρινό και το προσεχές πρόγραμμα εργασίας προβλέπουν για το Ινστιτούτο την διεξαγωγή ποικίλων δράσεων για την καταπολέμηση των στερεοτύπων ξεκινώντας από τη συλλογή πληροφοριών για τον τρόπο με τον οποίο οι άνδρες και οι γυναίκε παρουσιάζονται στα μέσα μαζικής ενημέρωση, αλλά και για τις πρωτοβουλίε ευαισθητοποίηση ως προς ε, τους ε, ρόλους προτύπου για τον άνδρα και τη γυναίκα, τους ακριβώ να καταπολεμήσουμε τα στερεότυπα. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Ξανά ο λόγο στην κυρία Λιωτάρ για να τελειώσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ε, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους έκαναν και όλες όσες έκαναν σχόλια. Έχουμε πολύ υλικό πλέον. Άκουσα πολύ προσεκτικά όλα όσα είπαν οι συνάδελφοι μία συνάδελφος ιδιαίτερα επέκρινε αρκετά σημεία της έκθεσης, θα συζητήσω μαζί της και προσωπικά. Οι γυναίκες, είπε, θέλουν ευέλικτες θέσεις εργασίας. Οπότε η ερώτησή μου είναι η εξής. Γιατί οι γυναίκες θέλουν ευέλικτες θέσεις εργασίας? Γιατί θέλουν οι ίδιες να ασχολούνται με τα παιδιά τους. Οκ, αν είναι έτσι δεν έχω κανένα πρόβλημα. Σε άλλες περιπτώσεις όμως οι γυναίκες κάνουν αυτή την επιλογή επειδή αυτό αντιστοιχεί σε, στην εικόνα που επιβάλλει η κοινωνία. Αν μια γυναίκα δεν ασχολείται με τα παιδιά της θεωρείται κακή μητέρα πολλές φορές. Απ' την άλλη μεριά υπάρχουν και πατεράδες οι οποίοι θα ήθελαν ευέλικτη θέση εργασίας, ευέλικτη εργασία για να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στα παιδιά τους. Οπότε πράγματι υπάρχει ένα πρόβλημα. Αν εξακολουθεί να υφίσταται αυτή η εικόνα στην κοινωνία, στην έκθεσή μου προσπαθώ να πω όχι ότι οι νέες γυναίκες δεν θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την ευελιξία υπάρχει ένα φαινόμενο το οποίο ε, χαρακτηρίζει την κοινωνία μας και πολλές φορές οι γυναίκες κάνουν αυτή την επιλογή ακριβώς για να ε, ε, σεβαστούν αυτό το μοντέλο για να μείνουν μέσα στα πλαίσια αυτού του μοντέλου. Τώρα, για τις σταδιοδρομίες, πυροσβέστες, για παράδειγμα. Στις κάτω χώρες η, λέξη για τους πυροσβέστες είναι μόνο στο αρσενικό γένος. Ε, στα Ολλανδικά η λέξη πυροσβέστης είναι άντρας της φωτιάς. Έτσι λέγεται. Και αυτό είναι ανησυχητικό. Και η νέοι από πολύ μικροί θα πρέπει να καταλάβουν ότι δεν θα πρέπει κάποιος να θεωρείται ε, εκεντρικός ε, αν θέλει να γίνει νοσοκόμος ένα αγόρι και το αντίθετο για τις γυναίκες. Ε, για τους δείκτες, ναι, συμφωνώ θα πρέπει να έχουμε δείκτες ε, για να μετράμε την πραγματικότητα. Το τι είδους δείκτες θα πρέπει να το σκεφτούμε Ένα άλλο συνάδελφο, μία άλλη συνάδελφο, είπε ότι η ευαισθητοποίηση είναι ένα πολύ καλό εργαλείο, συμφωνώ απόλυτα. Μετά προς την Κομισιόν θέλω να πω το εξής. Χαίρομαι που ασχολείστε με αυτό το ζήτημα σε διάφορα επίπεδα. Γνωρίζω ότι η Κομισιόν εργάζεται ε, επιμόνως για αυτό το ζήτημα, αλλά λυπάμαι που δεν έχει ενταχθεί το θέμα αυτό σε όλες τις δραστηριότητε της Κομισιόν. Πριν από ένα χρόνο έθεσα σε όλες τις γενικές διευθύνσει της Κομισιόν ε, το ερώτημα τα τελευταία πέντε χρόνια στο πρόγραμμα εργασία σα, ποια είναι, ποιες είναι οι δράσεις που οποίες είχατε αναλάβει, ποιες είναι οι προτάσεις που είχατε κάνει για την καταπολέμηση των στερεοτύπων των σχετικών με το φύλλο. Και μπορώ να σας ε, ομολογήσω ότι το αποτέλεσμα ήταν εξαιρετικά απογοητευτικό. Το άλλο ερώτημα που είχα θέσει ήταν τι πρωτοβουλίες σκοπεύετε να αναλάβετε τα επόμενα πέντε χρόνια. Και πάλι δεν πήρα καμία απάντηση στην πραγματικότητα. Σε όλα τα επίπεδα όμως, ε, στην κοινωνία, στην οικονομία, στην ε, επιστημονική έρευνα, στην καινοτομία, θα πρέπει να δράσουμε παντού. Μια γενική διεύθυνση μπορεί ασφαλώ να αρπάξει τον τάβρο από τα κέρατα, αλλά αυτό δεν αρκεί. Χρειάζονται και οι υπόλοιπε γενικέ διευθύνσει να ακολουθήσουν. Θα ήθελα λοιπόν να καλέσω την Κομισιόν, ε, την εκπρόσωπο της Κομισιόν εδώ, να περάσει αυτό το μήνυμα και στις άλλες γενικές διευθύνσεις. Σας ευχαριστώ. Και θα ήθελα να υπογραμμίσω πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα. Γιατί εδώ ουσιαστικά μιλάμε για την, ε, τις ευκαιρίες που θα έχουν τα παιδιά αυτά, κορίτσια, αγόρια, στις ζωές τους. Γιατί να τους δώσουμε μισές ευκαιρίες, να έχουν 100% της επιλογής από όλο το φάσμα επαγγελμάτων που ε, ήταν ικανά να ε, κάνουν. Τα στερεότυπα ξέρουμε ότι κλείνουν το δρόμο, δεν αφήνουν τον άνθρωπο να δουλέψει όπως θα ήθελε, να κάνει τη ζωή του όπως θα την ήθελε, γιατί επηρεάζει τις επιλογές του τελικά το στερεότυπο. Γι' αυτό πρέπει και να κοιτάξουμε αυτή την επίδραση και τα όρια όπου βρίσκονται αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν για αυτή τη δουλειά και θα ήθελα να σας ενημερώσω για το χρονοδιάγραμμα. Η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών είναι 18 Σεπτεμβρίου και η συζήτηση των τροπολογιών θα γίνει στις 10 Οκτωβρίου στην Επιτροπή μας. Η δε ψηφοφορία προβλέπεται για την Επιτροπή στις 6 Νοεμβρίου και στην Ολομέλεια ε, του Δεκεμβρίου, μάλλον θα δούμε το θέμα αυτό. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ για τη συζήτηση και πάμε στο σημείο 10 της ημερησίας διατάξεως που αφορά το πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 2014-2020 και δίνω το λόγο στην κυρία Γιανακουδάκη. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. θα ήθελα να εκφράσω την, ε, τον μεγάλο ενθουσιασμό με τον οποίο ανέλαβα αυτή την ε, έκθεση, γιατί όπως πάντα στα θέματα των γυναικών αισθάνεται κανείς ότι μπορεί να αλλάξει κάτι. Αν και πρέπει να σας πω ότι κατόπιν ε, μελέτης πιστώνω ότι λίγα πράγματα μπορώ να αλλάξω και θα ήθελα γι' αυτό να σας εξηγήσω από πού ξεκινάμε και μέχρι πού μπορούμε να πάμε. Ε, γιατί πρέπει να πω ότι ήμουν, ξεκίνησα με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό, αλλά τα φτερά μου σιγά σιγά κόπηκαν και η γραμματεία της Επιτροπής Βεβαίω προσπάθησε να περιορίσει την ε, άνοιξή μου, την όρεξή μου για ε, αλλαγές. Λοιπόν, έχουμε την αλλαγή του προγράμματος, να δούμε πώς ε, προχωράει. Δεν μπορούμε εμείς να μιλήσουμε για αύξηση των κονδυλίων, αλλά περισσότερο να συζητήσουμε το πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε προσθέμενη αξία για τις γυναίκες, από την άποψη δηλαδή της Επιτροπής μας. Άρα αυτά είναι τα όρια που ε, αντιμετωπίζουμε για την έκθεση αυτή. Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα βεβαίως για τις γυναίκες είναι η χρηματοδότηση Καλό αυτό, αλλά το κακό είναι ότι δεν μπορούμε να κοιτάξουμε τη μικροχρηματοδότηση, δηλαδή κάτω από τι 150.000, άρα δεν ασχολείται πραγματικά με τι ε, μικρομεσαίες επιχειρήσει, αλλά αυτό το παρουσίασα στην εξήγησή μου, στην αιτιολόγηση. Ίσως λοιπόν αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε με την έκθεσή μου θα ήταν να ενισχύσουμε τους τομείς ε, της χειραφέτησης μέσω της κατάρτισης και να ενθαρρύνουμε τις γυναίκες να κοιτάξουν ε, διαφορετικές επιλογές επιχειρηματικές που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες. Και κάτι ακόμη το οποίο έχουν σωματώσει, πρέπει να πω ότι μου εξήγησε η γραμματεία ότι δεν είναι δυνατόν στην πράξη να υλοποιηθεί, άρα θα πρέπει να βρούμε μια πρακτική λύση, είναι η ανάγκη να συγκεντρώνονται περισσότερα δεδομένα για το τι ακριβώς κάνουν οι γυναίκε και σε ποιου τομεί δραστηριοποιούνται και για να εντοπίζουμε έτσι πού μπορούμε και πού χρειάζεται να βοηθούμε. Ε, άρα σε αυτό το θέμα ίσως χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια και συντονισμός. Δεν είχα την ευκαιρία να συζητήσω με τους εισηγητές, λέει ο Μιλήτρια, και έτσι περιμένω να ακούσω τις δικές σας απόψεις για να προσδορίσουμε το χρονοδιάγραμμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κλάς έχει το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ και ευχαριστώ την κυρία Γιαννεκδάκη για την πολύ καλά ισορροπημένη έκθεση. Έχει επιλέξει μια πολύ καλή προσέγγιση και η έκθεση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να σα πω ήταν καλή και ισορροπημένη. βεβαίω θέλουμε να τη βελτιώσουμε στο βαθμό του δυνατού και ακριβώ σε αυτό θα επιμείνουμε στα θέματα στα οποία έθεσε το δάκτυλο του Δίπον των συνάδελφος. Δηλαδή, δεν έχουμε μόνο να κάνουμε οικονομικά ζητήματα που βεβαίω πλήττουν και ενώ και δεδομένης οικονομικής κρίσης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις γυναίκες. Αλλά έχουμε να κάνουμε και με τη γύρενση του πληθυσμού, δηλαδή τις δημογραφικές εξελίξεις ε, που παρατηρούνται και το γεγονός ότι έχουμε λιγότερο εργατικό δυναμικό στη θέσή μας μικρότερο πληθυσμό γενικότερα. Άρα αυτό πρέπει να το ενσωματώσουμε στη θεώρηση. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις συμβάλλουν τα μάλα στην οικονομία της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολύ σωστά δίνει στοιχεία μιλώντας για 67% των θέσεων εργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη που εξασφαλίζουν οι μικρομεσαίες ε, επιχειρήσεις. Και άρα είναι προφανές ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία η δραστηριοποίηση αυτών των επιχειρήσεων με την προσφορά εργασίας που εξασφαλίζουν και εγώ ε, πρέπει να σας πω καθώς και η ιδιαίτερη μου πατρίδα είναι μια περιοχή της Υπέθρου ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία για την Υπέθρου για τα μικρομεσαία επιχειρήση γιατί δεν είναι συγκεντρωμένα στα αστικά κέντρα αλλά στα, στην ε, περιφέρεια περισσότερο και ιδιαίτερω έχουν σημασία για την προσφορά εργασία στις γυναίκες οι οποίες μπορούν έτσι και να δραστηριοποιηθούν αλλά και να χειραφερθούν τεράστια λοιπόν η προσφορά τους και την υποστηρίζουμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν προσπαθεί να εξασφαλίσει καλύτερες συνθήκες πλαισίου για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, πρόσβαση στα μέσα χρηματοδότησης και τις αγορές γενικότερα και ιδιαίτερες ομάδες στόχων που ορίζει βεβαίως, συμπεριλαμβάνουν και τις γυναίκες, οποίες πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη υποστήριξη. Στα όσα συζητήθηκαν μέχρι τώρα. Τα στερεότυπα, παραδείγματο προ το ρόλο των φίλων. Πρέπει να σα πω ότι και στην συζήτηση για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει παρισφρίουν πάντα είναι πιο επιφυλακτικό ένα ε, τραπεζίτη Φερρυπίν όταν πάει μια γυναίκα να του ζητήσει χρηματοδότηση, ένα κεφάλαιο εκκίνηση για να στήσει μια επιχείρηση. Είναι διαφορετική η αντιμετώπιση του όταν έχει έναν άντρα απέναντί του, ο οποίο έρχεται και του παρουσιάζει ένα επιχειρηματικό ε, σχέδιο. Άρα λοιπόν νομίζω ότι με την Επιτροπή Βιομηχανίας μπορούμε να έχουμε πολύ καλή ε, συνεργασία γιατί έχει την ε, καθήλυν ε, αρμοδιότητα, έχει την κυρία έκθεση δηλαδή αναλάβει. μπορούμε να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στις ομάδες στόχους και δι' τις γυναίκες εδώ, εμείς από πλευράς μας. Είμαι πολύ ευχαριστημένη από τις 11 τροπολογίες κυρίας Γιανακουδάκη με τις οποίες υπογραμμίζεται ιδιαίτερα των αναγκών των νέων ανθρώπων και των γυναικών. Συνδυάζει δηλαδή τη νεολαία με τις γυναίκες με ιδιαίτερη έμφαση. Και την πτυχή βέβαια της ισότιμης, της ισότιμης μεταχείρισης. Επίσης θα ήθελα να υποστηρίξω την απέτηση για καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοοικονομικά, χρηματοδοτικά μέσα, αλλά και σε προγράμματα κατάρτισης. Στο αυτό σημείο θα ήθελα και εγώ να καταθέσω μια τροπολογία για την ε, ε, κατάρτιση ε, και προαγωγή της χρήσης των ηλεκτρονικών μέσων, της κοινωνίας πληροφορίας δηλαδή και των γλωσσών τις, γνω... τις γλωσσικές γνώσεις θα πρέπει να υποστηρίξουμε. Διότι έτσι μπορεί η γυναίκα να βρει ευκαιρίες και, από... και στη διεθνή αγορά. Οι μικρές και μεσές επιχειρήσεις ε, πολύ συχνά αναπτύσσουν δραστηριότητες υπερσυνοριακά, ακόμη και στην παγκόσμια σκηνή. Άλλωστε αυτό το καθιστά δυνατέων το ίδιο το ίντερνετ. Όταν όμως δεν υπάρχουν υποδομές για την ανάπτυξη της δραστηριοποίησης στο εξωτερικό, τι θα γίνει. Και γι' αυτό θα ήθελα να πω ότι παραμένει το πρόβλημα της ε, πληροφορίας, των αυτοκινητοδρόμων της πληροφορίας που δεν έχουμε, των υποδομών αυτών που δεν έχουμε. Δεν έχουμε υποδομές, δεν έχουμε πολλές φορές εξ αυτού του λόγου και το θάρρος από πλευράς της γυναίκας ή το κίνητρο εκ μέρους της γυναίκας, δεύτερα στην ε, περιφέρεια, να αναλάβει μια πρωτοβουλία για μικρή και μεσαία επιχείρηση. Άρα βρισκόμαστε μέσα σε ένα κύκλο πάντα. Γυρνάμε γύρω-γύρω. Δεν υπάρχει υποδομή, δεν υπάρχουν υποδομές. Ε, είναι μακρύς ο δρόμος μέχρι το χώρο εργασίας ε, και άρα και η γυναίκα ε, μερικές φορές αναγκάζεται εκ των πραγμάτων να ιδρύσει δική της επιχείρηση, και ενδεχομένω να προσλάβει έναν δύο υπαλλήλου και με τη μικρομεσαία επιχείρηση θεωρεί ότι μπορεί να είναι πιο ανεξάρτητη, πιο, να ορίζει μόνη τη το χρόνο εργασία τη και έτσι να συνδυάσει αυτή την εργασία με την ίδρυση μια οικογένεια με τον οικογενειακό τη βίο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι αυτά τα πράγματα θα πρέπει να τα συζητήσουμε. Αυτή την εβδομάδα θα καταθέσω προτάσει που έχουν να κάνουν όχι μόνο με την υποδέστερη, τη μειονεκτική θέση που μπορεί να έχει η γυναίκα στον χώρο τη περιφέρεια, αλλά και το ιδιαίτερο δυναμικό που μπορεί να προσφέρει η γυναίκα ή που μπορεί να προσφέρεται καλύτερα στη γυναίκα, που πρέπει να αξιοποιήσουμε, γιατί ε, οι δημογραφικές πιέσεις μας αναγκάζουν να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατότητα, κάθε άνθρωπο, πάνω απ' όλα κάθε γυναίκα, γιατί υπάρχουν πολλές δυνατότητες, αλλά πρέπει να τις βοηθήσουμε να προχωρήσουν βήμα το βήμα, ως προς την χειραφέτηση, ως προς την ανεξάρτητη δράση, γιατί μην ξεχνάμε ότι όταν μια γυναίκα πάει να ζητήσει ακόμη και 5.000 ευρώ κεφάλαιο εκείνης από μια τράπεζα, θα βρει μπροστά της έναν άντρα ε, τραπεζίτη, ο οποίος θα της απορρίψει την πρόταση. Ε, ούτε καν θα την εξετάσει. Καλά, καλά. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει η γυναίκα να ξέρει ότι μπορεί να πάει μέχρι την τράπεζα, μπορεί να ζητήσει το κεφάλαιο κίνηση, μπορεί να εξασφαλίσει ένα ε, δάνειο, μπορεί να αναχρηματοδοτήσει στη συνέχεια περαιτέρω επενδύσει και έτσι να ξέρει βήμα το βήμα ότι μπορεί να έχει διαφορετικές επιλογές. Οι υποδομές λοιπόν που λείπουν, η πρόσβαση στις αγορές ε, είναι πολύ σημαντικά ζητήματα πρέπει από την οπτική γωνία των γυναικών να τα εξετάσουμε και να τα δούμε όχι μόνο σαν ε, ε, αρνητική διάκριση, αλλά και σαν μια δυνατότητα για θετική υποστήριξη για τις γυναίκες. Αυτά λοιπόν, πολλά σημεία, πολλά σημεία συζήτησης έχει αυτή, αυτό το θέμα. Ένα θέμα το οποίο πιστεύω μπορούμε από κοινού μας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επεξεργαστούμε έτσι ώστε να προχωρήσουμε καλά, με καλά αποτελέσματα, με ουσιαστικές ε, απτές και αποτελεσματικές τροπολογίες εγκαίρως. Ευχαριστώ και πάλι την εισηγήτρια για την πολύ καλή της έκθεση και τις τροπολογίες που έχει ήδη υποβάλει. Ευχαριστώ πολύ κυρία Παπαδοπούλου. Uh, Ευχαριστώ πρόεδρε. Συγχαίρω και εγώ την Μαρίνα Γιανακουδάκη για τις προτάσεις της. Πρόκειται για μια έκθεση που έχει πολλούς στόχους. Το νέο πρόγραμμα στοχεύει κυρίως ε, τους, ε, τις επιχειρηματίες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα ωφεληθούν από την μεγάλη ευκολότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση και ε, Επίσης ε, στοχεύει τους ε, ανθρώπους που θέλουν να λειτουργήσουν ως ελεύθεροι επαγγελματίες και αντιμετωπίζουν προβλήματα. Επίσης στοχεύει στο να βοηθήσει τις αρχές των κρατών μελών προκειμένου να ε, σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια πολιτική μεταρρύθμιση. Οι γυναίκες επιχειρηματίες είναι λίγες. Και αν δούμε τη σύγκριση των στατικών στοιχείων θα διαπιστώσουμε ότι πολλές γυναίκες στο νότο της Ευρώπης αλλά και σε πολλές άλλες ε, χώρες διστάζουν να ξεκινήσουν μια δική τους επιχείρηση και χρειάζονται πολύ ενθάρρυνση. Θα πρέπει και πάλι να αντιμετωπίσουν στερεότυπα, δεν έχουν τεχνογνωσία, δεν γνωρίζουν πώς μπορούν να έχουν εύκολη πρόσβαση στη χρηματοδότηση και αυτό θα πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε εμείς ως Επιτροπή ε, Γυναικών. παρόλο ότι υφίστανται πολλοί περιορισμοί, δεν μπορούμε να κάνουμε τα πάντα, δεν μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να προσθέσουμε κάποια αξία στη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να βοηθήσουμε τις γυναίκες ε, να... Ε, ξεκινήσουν δραστηριότητες που χρειάζονται επιχειρηματικό πνεύμα, επιχειρηματικές ικανότητες και να τους δώσουμε αυτές τις ικανότητες θα πρέπει να καταλάβουν πώ μπορούν να ξεκινήσουν τι δικέ τους επιχειρήσεις, πώς μπορούν να τι αναπτύξουν, πώ ε, θα βελτιώσουν την αυτοπεποίθησή του και να αλλάξουν και την ίδια του την οτροπία και τι αντιλήψει του. Χρειάζονται πολλή ενθάρρυνση. Θα πρέπει να στοχεύσουμε και τι ε, νέε γυναίκε, του νέου γενικότερα, όσο και τι ε, γυναίκες που σήμερα αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα στην εξασφάλιση των μέσων της χρηματοδότηση και της τεχνογνωσίας για να ξεκινήσουν δικές τους επιχειρήσεις. Ε, αναμένουμε ανυπομονησία να δω τους άλλους σκιώδεις ηγητές και την εισηγήτρια προκειμένου να το συζητήσουμε και να υποβάλουμε τις τροπολογίες που χρειάζονται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ως σκιώδης συγητής θα ήθελα να πω και εγώ το εξής. Η ε, κυρία Γιανακουδάκη έχετε συμπεριλάβει την διάσταση της ισότητας των φύλων ε, σε αυτή σας την έκθεση και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι ε, θα είναι πολύ καλή η γνωμοδότηση αυτή. Έχω όμως δύο σχόλια να κάνω. Πρώτον, η τροπολογία υπαριθμών 1. Δεν καταλαβαίνω γιατί διαγράψατε την οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και αποδοτικής χρήσης των πόρων και της ενέργειας. Τα αντικαταστήσατε όλα αυτά από τη φράση τόσο για, τους, για, τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άντρες. Νομίζω ότι είναι αρκετά εύκολο να ε, τα συμπεριλάβουμε και τα δύο. Δεν ε, αντιβαίνει το ένα στο άλλο θα μπορούσατε να διατηρήσετε αυτό που υπήρχε και ταυτόχρονα να προσθέσετε το, τόσο για τις άνδρες όσο και για τις γυναίκες. Ε, μετά, δεύτερο σχόλιο, ε, σε σχέση με την πρόταση της Κομισιόν αλλά και γενικότερα. Όταν μιλάμε για μικρομεσαίες επιχειρήσεις πιστεύω ότι μερικές φορές υπάρχει η τάση να δημιουργούμε έτσι μια φούσκα για το πόσο σημαντικά είναι όλα αυτά τα πράγματα. Είναι σημαντικά, αλλά πολλές φορές ξεχνάμε ότι τι είναι αυτό που μας οδηγεί, που μας διευκολύνει στο να ε, δημιουργήσουμε επιχειρήσεις, ε, να εξασφαλίσουμε ανάπτυξη και πρέπει να το δούμε πιο γενικότερα. Δηλαδή, οι γυναίκες θα πρέπει να διευκολυνθούν στο να συμμετέχουν στην οικονομία. Αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να έχουμε την απαραίτητη κοινωνική υποδομή. Για παράδειγμα, παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, βέβαια επίσης φροντίδες ε, για τους ηλικιωμένους. Αν δεν υπάρχουν αυτές οι υποδομές, τότε ποιος θα αναλάβει αυτές τις φροντίδες. Αυτές οι φροντίδες θα πρέπει να δίνονται στα παιδιά και στους ηλικιωμένους στο σπίτι, οπότε η γυναίκα δεν θα είναι ελεύθερη. Συνεπώς, ζητούμε καλύτερο ρόλο για τις γυναίκες, αλλά θα πρέπει να τις βοηθήσουμε πρακτικά. γνωρίζω πως ε, δεν μπορούμε να ζητάμε πράγματα σαν να ζητάμε δώρα από τον Άγιο Βασίλη. Αλλά για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό, ζωτική σημασία. Οι κοινωνικέ υποδομέ. Η συμμετοχή δεν αφορά μόνο τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, αλλά γενικότερα τη διευκόλυνση των γυναικών να συμμετάσχουν στην οικονομική ζωή. Αυτά ήθελα να πω. Θα δώσω το λόγο στην εκπρόσωπο τη Κομισιόν, αν επιθυμεί να μιλήσει. Η κυρία Μίτσελ. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια, καθώς επίσης και όλους τους βουλευτές που υπέβαλαν παρατηρήσεις. Αρχικά θα ήθελα να πω ότι δεν έχουμε καμία πρόθεση να περιορίσουμε τις φιλοδοξίες σας. Απλώς πρέπει να παραμείνουμε ρεαλιστές καθώς στοχεύουμε ψηλά. Συμφωνούμε απόλυτα με τους στόχους που εκφράζονται στην έκθεση και σε κάθε περίπτωση ως ε, γυναίκα που προσπάθησε σε ορισμένες περιπτώσεις να ξεκινήσει επιχειρηματική δράση, δεν θα μπορούσα παρά να συμφωνώ απόλυτα με τις ανησυχίες που εκφράζονται εδώ πέρα. Πολύ σωστά η κυρία Γιανακουδάκη μας λέει ότι ε, εξετάζουμε αυτή τη στιγμή ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και επομένως θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε σχέση με το τι μπορούμε να διευθετήσουμε και να συζητήσουμε στα πλαίσια του προγράμματος αυτού. Γενικότερα όμως όσον αφορά το ζήτημα των γυναικών επιχειρηματιών, Εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση της υποστήριξής τους. Μάλιστα πρόσφατα έχουμε και μία έρευνα η οποία συγκρίνει τα επίπεδα επιχειρηματικότητας στις γυναίκες ανάμεσα στη Βρετανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ορισμένοι θα περίμεναν ότι θα υπήρχαν κάποιες πολιτιστικές ομοιότητες, καθότι δεν υπάρχει καν διαφορά γλώσσας ανάμεσα στις δύο χώρες. Παρ' όλα αυτά η διαφορά είναι τεράστια. Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας, μια τεράστια απόσταση ουσιαστικά που χωρίζει τις ε, δύο αυτές χώρες θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μα τα όσα λέγονται για τις γυναίκες στην Ήπεθρο, για τις γυναίκες που πλήττονται από κοινωνικά στερεότυπα. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις δυσχέρειες. Όσον αφορά το πρόγραμμα COSME, τονίζεται στην έκθεση ότι αποτελεί τη συνέχεια του ΣΥΠ Το μόνο πρόβλημα που έχουμε με τη σχετική τροπολογία είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να συλλέξουμε όλα αυτά τα δεδομένα για τους δείκτες που απαιτείται από εμά. Που απαιτούνται, με συγχωρείτε, από εμά. Προφανώς ε, θέλουμε να κάνουμε ό,τι το δυνατό, αλλά πολλές φορές δεν γίνεται να καλύψουμε στόχους οι οποίοι είναι εκφύση αδύνατον να ικανοποιηθούν. Στα σημεία 9 και 13, στροπολογίες 9 και 13, δεν ξέρω καν αν τα δεδομένα αυτά υφίστανται και ακόμα και αν υφίστανται θα είναι μόνο σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο και ουσιαστικά δεν θα είναι συγκρίσιμα τα δεδομένα αυτά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν είμαι πεπισμένη επίσης ότι τα δεδομένα αυτά θα είναι τελικά αξιόπιστα και ότι μπορούν να συλλεχθούν σε τακτική χρονική βάση. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση, θα ήθελα απλώς να τονίσω ότι υπάρχει ακόμα η δυνατότητα της μικροχρηματοδότησης στα πλαίσια του κόσμου μέσω του συστήματος εγγύσεων. Η επιλογή της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, είναι συνειδητή. Προτείνουμε ένα πρόγραμμα καινοτομία, το οποίο συμπεριλαμβάνει ουσιαστικά τη συνιστότητα τη χρηματοδότηση. Επομένω, υπάρχει δυνατότητα μικροχρηματοδότηση, απλώ δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε εδώ πέρα επικάλυψη. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μα, επομένω δεν θα επισέλθω σε πολλέ λεπτομέρειε. Ωστόσο, θα ήθελα να τονίσω ότι ε, στα μέσα Οκτωβρίου θα έχουμε μία σύνοδο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μία μέρα ουσιαστικά η οποία θα αφιερωθεί στις γυναίκες που δραστηριοποιούνται στα πλαίσια των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων και είμαι σίγουρη ότι θα δω πολλά γνωστά πρόσωπα να συμμετέχουν στα διάφορα πάνελ και σε ομάδες εργασίας. Ως πρόγευση, με την άδεια μάλιστα του Προέδρου, μπορώ να σας αφήσω κάποια αντίτυπα τα οποία μόλις εκτυπώθηκαν όσον αφορά το μυστικό της επιτυχίας για τις μικρομισές επιχειρήσεις σε διεθνές επίπεδο, ένα ζήτημα το οποίο αντιμετωπίσαμε και στο παρελθόν, όπου βλέπουμε, θα δείτε στα έγγραφα αυτά και στα παραδείγματα που δίνουμε, ότι ε, τουλάχιστον το 50% των ε, επιχειρηματιών στις περιπτώσεις αυτές είναι γυναίκες. Όχι μόνο στον τομέα των τροφίμων και της μόδας, αλλά πολλές φορές ακόμα και της ναυπηγίας, του περιβαλλοντικού ελέγχου ή ακόμα και των υπηρεσιών ασφαλείας ή ακόμα και γυναίκες που στείλουν επιχειρήσεις στον τομέα της ξυλουργίας και των σχετικών υποδομών. Επομένως θεωρώ ότι ε, το έγγραφο αυτό πραγματικά περιλαμβάνει κάποια πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Είμαστε στη διάθεσή σας και για τις τροπολογίες βέβαια που θα ε, υποβληθούν και για τις υπόλοιπες λεπτομέρειες που θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και στο μέλλον όσον αφορά την έκθεση αυτή, Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Γιάννη Κουδάκη, έχετε το λόγο. <laughs> no way. <laughs> I'll deal with you last. <laughs> Όχι, εσάς σας αφήσω για το τέλος. Το αγαπημένο μου τραγούδι είναι αυτό που λέει «Μπορώ να πετάξω, I can fly» και άρα μη μου λέτε τι δεν μπορώ να κάνω. Εν πάση περιπτώσει όμως, αυτά που λέτε ενισχύουν ε, την διαπίστωση ότι η έκθεση αυτή έχει περιορισμούς, έχει όρια, με βάση αυτά θα εργαστούμε. Θα τα καταφέρουμε όμως, άλλωστε ιστορία εδώ γυναίκες είμαστε. Λοιπόν, αντιλαμβάνομαι ποια είναι τα προβλήματα, αντιλαμβάνομαι επίση ότι πρέπει να κοιτάξουμε κάποια πράγματα, πώς μπορούμε δηλαδή τα προβλήματα να τα περιορίσουμε. Περιμένω να ακούσω προτάσεις, τροπολογίες. Περιμένω να δω τις τροπολογίες. Ήδη ήταν ενδιαφέρουσες και από τις δύο πλευρές οι υποδείξεις. Ως επιχειρηματίας, επιχειρηματίας δεν πρέπει να πω ότι όσο πιο πολλές διαφορετικές είναι οι γωνίες από τις οποίες έρχονται οι προτάσεις, τόσο πιο πλούσια μπορεί να γίνει η δουλειά, τόσο πιο καλή η έκθεση. Τώρα, ε, αν μπορούμε να έχουμε βρεφονιπιακούς σταθμού και αν θα πρέπει αυτού να του πληρώνουν ε, οι μικρομεσαίε επιχειρήσει, ή αν θα πρέπει να του ιδρύσει το κράτο και πίσω να τους χρηματοδοτεί, δεν είναι η ώρα μάλλον να την κάνουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει περιμένω πότε θα έρθει η ώρα να τη συζητήσουμε. Και σα ευχαριστώ πολύ που ήσασταν όλοι εδώ σήμερα για τη συζήτηση. Ο Πρόεδρος, βεβαίως, βεβαίως, και εγώ περιμένω με αδημονία τη συζήτηση αυτή. Σας ευχαριστώ για τη συζήτηση. και θα ήθελα να μου επιτρέπετε να ανακοινώσω κάποιες πληροφορίες για το χρονοδιάγραμμα της γνωμοδότησης προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών στην γνωμοδότηση της κυρίας Γιανακιουδάκη είναι η 30 Αυγούστου, 30 Αυγούστου, ψηφοφορία στην Επιτροπή μας 19 ή 20 Σεπτεμβρίου και η Επιτροπή Βιομηχανίας θα επιληφθεί 8 και 9 Οκτωβρίου για να πάμε στην Ολομέλεια στη δεύτερη μηνή ολομέλεια, στη δεύτερη ολομέλεια του Νοεμβρίου, λέει τη μήνυ ολομέλεια. Και τώρα κλείσαμε το θέμα αυτό και περνάμε στο 11, Γενικό Προπολογισμό Ευρωπαϊκή Ένωση για το Οικονομικό έτο 2013, όλα τα τμήματα. Μα πιέζει πολύ ο χρόνο και έτσι παρακαλώ την εισηγήτρια, κυρία Χάνιμπολ, να λάβει το λόγο αμέσω. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα είδατε, φαντάζομαι, τι τροπολογίε που κατατέθηκαν. Είναι πολύ απογοητευτική η κατάσταση. Πρέπει να πω ότι δεν μας ξαφνιάζει το ότι προσπαθεί το Συμβούλιο να περικόψει τις αυξήσεις που εμείς προτείναμε. Αλλά ακόμη και με το υφιστάμενο οικονομικό κλίμα δεν στέκουν αυτά που προτείνει, γιατί είναι πολύ σημαντικές οι γραμμές που πάει να περικόψει το Συμβούλιο. Περιλαμβάνουν παραδείγματι τις συνθήκες εργασίας υπό, υπό τον τίτλο «Απασχόληση κοινωνική αλληλεγγύη ισότιμη μεταχείριση» με 14,84% προσπαθεί να περικόψει το Συμβούλιο στην κοινωνική ανάπτυξη και πρόοδο 22% περικοπό, περικοπή, ισότητα των φύλων στο Ινστιτούτο για, την ισότητα των φύλων 4% περικοπή, καταπίεση, καταπίεση βία, κοινωνική κατάρτιση 69%. 6,9% περικοπή και έτσι ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις πιέσεις, να βρούμε περισσότερη χρηματοδότηση για το πρόγραμμα Δάφνη, στο οποίο έχουμε πολύ μεγάλες πιέσεις και πρέπει να πω ότι βρίσκω καταθλιπτική όλη αυτή την κατάσταση. Αυτό που προτείνω λοιπόν είναι να μην υποχωρήσουμε σε αυτό το στάδιο, θα ήταν λάθος να υποχωρήσουμε, να εμείνουμε στα όσα θέλουμε, να καταφέρουμε να κάνουμε τροπολογίες με επαναφορά των ποσών, όπως τα είχαμε προσδιορίσει, και είναι παράδοξο κιόλα, γιατί αν κάνει κανείς τα, την άρθρηση θα δει ότι η επαναφορά των ποσών στις δεσμεύσεις του 2012 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνεπάγεται αύξηση για τον προϋπολογισμό στους τομείς αυτούς κατά 9,527,04 ε, ευρώ, δηλαδή ούτε καν 2% αύξηση. Και αυτό είναι που δεν καταλαβαίνω εδώ πέρα και γι' αυτό αισθάνομαι και τόσο μεγάλη απογοήτευση. Τι μπορεί κανείς να καταφέρει εάν περικοπούν αυτά τα ποσά, που είναι τόσο λίγο, τόσο λίγη περικοπή. Από την άλλη τα ποσά αυτά μπορούν να καταφέρουν τεράστιες, να επιφέρουν τεράστιες αλλαγές και πρόοδους. Γι' αυτό λοιπόν ζητούμε μια ελάχιστη αύξηση πολύ σημαντική για τις γυναίκες και την ισότητα των φίλων και επιμένω και προτείνω να μην ε, εγκαταλείψουμε τον αγώνα ακόμα. Όσον αφορά τα πιλωτικά προγράμματα είναι κάπως καλύτερη κατάσταση. Τέσσερα έχουμε προβάλλει προαγωγή των ε, γυναικών στον επαγγελματικό βίο και αναπροσαρμογή για πράσινες γυναίκες, για πράσινες θέσεις εργασίας, δίκτες για την ε, υλοποίηση της, του χάρτη ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, συνθήκες ισότητας μεταχείρισης κλπ. Οι τρεις πρώτες προτάσεις είχαν ε, κακές επιδόσεις. C και D βαθμολογία πήραν. Η τέταρτη όμως, δηλαδή η εφαρμογή του χάρτη ε, ισότητα μεταξύ των και γυναικών στο τοπικό επίπεδο είχε τον καλύτερο βαθμό α και άρα ίσως μπορούμε να περιμένουμε καλές, ε, καλή συνέχεια. Επομένως είχαμε ένα εκατομμύριο ευρώ. Δεν είναι βέβαιο ότι θα τα πάρουμε εν τέλει, αλλά πάντως ε, είναι σε καλό δρόμο αυτό το πρόγραμμα, αυτή η πιλωτική προσπάθεια. Καλή είδηση. Δεδομένου δεν είχαμε και ποτέ πιλωτικό έργο στο παρελθόν η Επιτροπή μας και ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε. Πολύ σύντομα λοιπόν να σας πω ακόμη δύο-τρία πράγματα. Ξέρω ότι πιέζει ο χρόνος. Αυτά που κάνει η Επιτροπή για να δώσει περισσότερη έμφαση στη προοπτική και τη διάσταση του φύλου, η προσπάθεια αυτή για ενσωμάτωση της δράσης του φύλου βεβαίω σε κάθε είδους πολιτική ε, φέρνει καρπούς. Η καταπολέμηση της ε, εγκληματικότητας έχει οδηγήσει μια τροποποίηση σχετικής ε, διατάξεως προκειμένου να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό της βίας ακόμη και σε περίπτωση στενών συγγενικών σχέσεων. Εκεί δηλαδή όπου έστω και αν ε, κινδυνεύουμε να χάσουμε την χρηματοδότηση από το Συμβούλιο έχουμε πολλές απαιτήσεις. Το 1936 έχουμε κάνει μια τροποποίηση για την ε, ενσωμάτωση της σημασίας της εξορρόπησης των φύλων εξωτερικές δράσεις και σημαντικά προγράμματα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, ασκεί την πολιτική αυτή και να την ασκεί ορατά η ίδια. Αυτό κάνουμε λοιπόν στο σημείο 44-448 υπάρχει επίσης η διάσταση του φύλου και η απασχόληση με ισοτιματικό που έχει αντιμετωπιστεί και υπό την πτυχή φύλλο, απασχόληση ανεξαρτητός φύλλου και προοπτικές, γιατί είναι πολλές οι γυναίκες οι οποίες βρίσκονται σε επισφαλή θέση εργασίας ή υπάρχουν παραδείγματι λεγόμενες ρόζο θέσεις εργασίας, ε, γυναικών δηλαδή ειδικά, που έχουν ε, περιορισμένα συμβόλαια ή πολύ ε, χαμηλές αποδοχές και λοιπά πλέον εκτήματα. Και φυσικά παραμένει πάντα το χάσμα το μισθολογικό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευθεί να το καλύψει. Μια στρατηγική ισότητα, ε, για την ε, ε, για τη σχέση μεταξύ ανδρών και γυναικών στο προσεχές διάστημα συμπεριλαμβάνει και το κλείσιμο αυτής της ψαλίδας. και άρα υπάρχει καλή πρόεδρε, πρόοδος, αλλά κύριε Πρόεδρε νομίζω ότι είναι απογοητευτικό το ότι ασκούνται τόσε πιέσει για τον περιορισμό τη χρηματοδότηση. Πάντω, εμεί θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε μέχρι το τέλο. Και θα ήθελα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ρωτήσω εάν, πρώτον, εφόσον περικοπεί ο προπολογισμό σε σχέση με τα ποσά του 2012, έχει η περικοπή αυτή στηριχθεί σε ενδεχόμενη μία απορρόφηση πόρων από το προηγούμενο έτος. Υπάρχει κάπου δηλαδή που μπορούμε να πούμε να, εδώ δεν δαπανήθηκαν τα κονδύλια, μπορούμε από εκεί να κάνουμε την περικοπή. Ή είναι τυχαίες και οριζόντιες οι περικοπές. Αυτή ήταν η πρώτη μου ερώτηση. Και η δεύτερη είναι γιατί είναι τόσο μεγάλες οι περικοπές ως προς το κομμάτι που αφορά το, την καταπολέμηση και την πρόληψη κλιματικότητας. 64.400.000 εκατομμύρια 400 ευρώ. Που ουσιαστικά διαγράφει όλη τη γραμμή του προπολογισμού. Επομένω, γιατί ένα τόσο σημαντικό θέμα έχει πω ήταν τόσο σημαντικό πλήγμα. Περιμένω από τι προτάσει και τι απαντήσει τη Επιτροπή. Ευχαριστώ. There's no member asking for the floor, but uh, I will just briefly say that. Ξαναγυρίζω στα σουηδικά. Θέλω απλώς να πω δύο πράγματα εν συντομία. Ε, συμμερίζομαι την ε, απογοήτευσή σας και συμφωνώ με τις τάσεις σας σε ό,τι αφορά το ρόλο μας ως Επιτροπής. Εμείς έχουμε την ευθύνη να μιλάμε για το τι χρειάζεται και να ζητούμε να καλυφθούν οι ελλείψεις προκειμένου να έχουμε μια αποτελεσματική πολιτική. Αυτή τη στιγμή το θέμα δεν είναι μόνο η οικονομική υπευθυνότητα, σε εισαγωγικά. Ο ρόλος μας είναι να εντοπίσουμε τις ανάγκες, να πούμε τι πιστεύουμε ότι χρειάζεται να γίνει με το πρόγραμμα Δάφνη, τι πρέπει να γίνει με τα όλα όσα σχετίζονται με τα δικαιώματα ανδρών και γυναικών και αργότερα άλλοι θα κρίνουν όλα αυτά από οικονομικής πλευράς. Αυτή τη στιγμή εμείς αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι να εντοπίσουμε τις ανάγκες. Οι ανάγκες λοιπόν υποδεικνύουν αύξηση της χρηματοδότησης των προγραμμάτων το πρόγραμμα Δάφνη είναι πολύ σημαντικό και σφαιρικό, αλλά θα πρέπει να το εξασφαλίσουμε επαρκή χρηματοδότηση. Συνεπώ, συμφωνώ μαζί σα ότι αυτή τη πρέπει να μιλήσουμε για τι ανάγκε. Τούτου λεχθέντο, θα δώσω το λόγο στην κυρία Κβατόρσκα. Ελπίζω να προέφερα σωστά το όνομά τη. Κυρία Κουαρτέσκα από την Κομισιόν, Ευχαριστώ που δίνετε το λόγο στην Κομισιόν, Πρόεδρε. Σε σχέση με την πρώτη ερώτηση για το πρόγραμμα Δάφνη. Ο, το προσχέδιο προπολισμού 2013 προτείνει 18 εκατομμύρια σε επιστώσεις ανάλυση υποχρεώσεων. Όμως στην πράξη αυτό αποτελεί μείωση σχέση με το 2012. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του προπολογισμού του 2012 η Δημοσιονομική Αρχή είχε αυξήσει τη χρηματοδότηση του 2012 κατά 2 εκατομμύρια στα 19,5 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε γι' αυτό λόγο βλέπουμε τη μείωση. Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη ερώτησή σας. Η μείωση σε σχέση με τον προπολογισμό του 2012 σε ό,τι αφορά τα κονδύλια, σε ό,τι αφορά την πρόταση της Κομισιόν για το προσχέδιο προπολογισμού του 2013 για τα προγράμματα Δάφνη, όπως επίσης και τις δύο πτυχές του Progress, εμείς προτείνουμε τα ίδια ποσά για το 2013 με αυτά που είχαμε προτείνει το 2012. Δεν προτείνουμε περικοπή. Αν δούμε και την επίδοση για το 2011 το ποσοστό υλοποίησης ξεπερνάει το 90% για όλα αυτά τα προγράμματα, το ποσοστό απορρόφησης. Ε, ε, Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Επιστρέφουμε στην εισηγήτρια. Κυρία Χάνιμπολ. Um, Ευχαριστώ για τις απαντήσεις. Συμφωνώ πλήρω με τα όσα είπε ο πρόεδρο προηγουμένω. Θα πρέπει να επιμείνουμε στην στάση μα. Η δική μα δουλειά είναι να εξασφαλίσουμε επαρκή χρηματοδότηση για τι γυναίκε και για την ισότητα των δύο φύλων. Αυτή είναι η αποστολή τη Επιτροπή μα. Δεν είναι δυνατόν να την απαρνηθούμε αυτή τη στιγμή. Και πράγματι, αυτή τη στιγμή ε, δεν έχουμε στο μυαλό μας το συνολικό προπολογισμό. Εμείς πολεμάμε αυτή τη στιγμή για να εξασφαλίσουμε το δικό μας μερίδιο. Δεν μιλούμε για τον προπολογισμό στο σύνολό του, για το κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επιφέρει μειώσει ή όχι. Εμείς απλώς πρέπει να εξασφαλίσουμε επαρκή χρηματοδότηση για τα δικαιώματα των γυναικών και για την ισότητα των δύο φύλων. Συνεπώ, θα ήθελα παρακαλώ πολύ να με υποστηρίξετε στην ομοδότησή μου. Tack så mycket eh, Πρόεδρος, σας ανακοινώνω το εξής. Η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι 26 Ιουλίου, 12 το μεσημέρι. Η Επιτροπή μας θα ψηφίσει στις 3 Σεπτεμβρίου και τον Οκτώβριο θα ψηφίσει η Επιτροπή Προπολογισμών. Τελειώσαμε και με αυτό το ζήτημα. Περνάμε στο 12. Έχουμε μείνει πίσω. Μας πιέζει ο χρόνος. Ε, γίνεται να το συζητήσουμε στα επόμενα τέσσερα λεπτά, κυρία συντάκτηρα της νομοδότησης. Ή θέλετε να το περιμένουμε το απόγευμα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομη. Νομίζω ότι τέσσερα λεπτά επαρκούν. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω λοιπόν την γνωμοδότησή μου όσον αφορά την συνοχή της συναπτυξιακής πολιτικής για το 2011. Βασική Επιτροπή εδώ είναι η Επιτροπή ανάπτυξη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Γραμματεία για την εξαιρετική συνεργασία που είχα μαζί τη. Είναι περιορισμένη η έκταση της γνωμοδότησης γιατί ήταν αδύνατο να συμπεριλάβω όλες τις παρατηρήσεις τις οποίες έλαβα. Προσπάθησα λοιπόν να επικεντρωθώ στο ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως όσον αφορά τις γυναίκες και τα κορίτσια στις αναπτυσσόμενες χώρες. Δεν θα αναφερθώ στην έκθεση της Επιτροπής. Φαντάζομαι ότι οι σκιώδεις ηγητές θα διαβάσουν από μόνοι τους αυτή την έκθεση. Στη γνωμοδότησή μου επικεντρώνομαι στα ζητήματα τα οποία θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικά γιατί άπτονται των θεμελιωδών δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών. Ο τομέας της ανάπτυξης συνδέεται στενά με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Επομένως, επικεντρώνομαι στο ζήτημα της υγείας των γυναικών και των παιδιών, ιδίω των νέων κοριτσιών και την βία κατά των γυναικών και των νέων κοριτσιών. Στις αναπτυσσόμενες ε, χώρες πολύ συχνά οι υποδομές κοινωνικής πρόνοιας είναι πολύ αδύναμες. Πολύ συχνά οι γυναίκες και τα κορίτσια δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στα απαραίτητα ανθρώπινα δημοκρατικά δικαιώματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τροποποιηθεί η νοοτροπία απέναντι στις γυναίκες και να σταματήσουν πλέον οι άντρε, τα αγόρια, να βρίσκονται, να έχουν την πιο ευνοϊκή μεταχείριση. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει η διαπαιδαγώγηση των πολιτών είναι τέτοια που να μπορούν να αποφεύγονται επίσης ε, οι ε, σεξουαλικές παρανοχλήσεις, η εκτεταμένη βία λόγω φύλου, καθώς επίσης και αναγκαστική γάμη. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να ενημερωθούν οι γυναίκες για την σεξουαλική και παραγωγική τους υγεία. Η ενημέρωση αυτή, η ευαισθητοποίηση αυτή αποτελεί βάση για την καταπολέμηση πολύ σημαντικών ασθενειών, θανατηφόρων ασθενειών όπως το AIDS και επίσης μπορεί να ενισχύσει γενικότερα τη θέση των γυναικών στην κοινωνία. Αυτό βασίζεται και στην πλατφόρμα Πεκίνο ΣΥΝ 15 δεν θα επαναλάβω τα όσα λέγονται στην πλατφόρμα αυτή. Είναι ένα ζήτημα το οποίο το συζητάμε πάρα πολύ συχνά στην Επιτροπή μας. Ο ορισμός που προβλέπεται στην πλατφόρμα αυτή δεν κάνει λόγο μόνο για την άμβλωση. Τα όσα λέγονται πάντω στο, στο εν λόγω σχέδιο δράση θα πρέπει να ισχύουν προφανώ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στι αναπτυσσόμενε χώρε. Όσον αφορά τώρα του βιασμού και την σεξουαλική βία, Πρόκειται για ένα φαινόμενο το οποίο επηρεάζει πάρα πολύ την ζωή των γυναικών. Δεν αποτελεί όμως φαινόμενο που περιορίζεται μόνο σε εμπόλεμες περιοχές. Υπάρχουν πολλές γυναίκες και κορίτσια που αντιμετωπίζουν γενικότερα φαινόμενα βίας, τα οποία έχουν να κάνουν με την οτροπία και τις παραδόσεις ορισμένων χωρών, όπως για παράδειγμα ο ακροτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων, το ότι υπάρχουν διάφορες πρακτικές προγενετικής επιλογής, ότι πολύ συχνά υπάρχουν φαινόμενα παιδοκτονίας θηλαίων βρεφών κτλ. Όλα αυτά αναφέρονται στο σημείο 2 της γνωμοδότησής μου. Θα ήθελα προφανώ να γνωρίζω ποια είναι η άποψη των αδέλφων μου. Δεν υπάρχει απαραίτητο χρόνος σήμερα. Πιστεύω πάντως ότι θα καταβάλλετε, καταθέσετε με συγχωρείτε Και θα ήθελα επίση να προσθέσω ότι τα δικαιώματα των γυναικών όσον αφορά την περιουσία, την ακίνητη περιουσία, αποτελεί επίσης ένα θεμελιώδες δικαίωμα. Θεμελιώδες όμως δικαίωμα το οποίο δεν μπόρεσα να συμπεριλάβω σε αυτή τη γνωμοδότηση. Προτίμησα, όπως είπα στην αρχή της παρεμβασής μου, να επικεντρωθώ σε κάποια άλλα σημεία. Ένα άλλο τομέα που δεν κατάφερα να συμπεριλάβω στην νομοδότησή μου είναι αυτό που έχει να κάνει με την αναγκαστική εργασία των παιδιών. Προσπάθησα, όπω εξήγησε, να επικεντρωθώ περισσότερα στα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών. Προσβλέπω σε τροπολογίε και σε περαιτέρω συζήτηση. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρο. Σα ευχαριστούμε. Όντω μα πιέζει πάρα πολύ ο χρόνο. Αν υπάρχει πάντως κάποιο ο οποίο θα ήθελε να πάρει τώρα το λόγο, Μάλλον ενδεχομένω καλύτερα να γίνει αυτό στο απόγευμα, μετά το μεσημεριανό διάλειμμα, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τον απαραίτητο χρόνο. Πρέπει να δώσω και τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρέμβει. Δεν ξέρω αν εκπρόσωπο Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να δώσουμε το απόγευμα. Πολύ σύντομα λοιπόν, α πάρει το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο πρόεδρο ευχαριστεί του διερμηνεί που θα παραμείνουν λίγο παραπάνω. Σα ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είμαι αρμόδια για τα ζητήματα συνοχής αναπτυξιακής πολιτικής. Δεν θα αναλώσω πάρα πολύ χρόνο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας που ασχολείται με την έκθεση αυτή, γιατί θα θέλαμε η, η έκθεση αυτή να συζητηθεί και εκτός Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να έχουμε πολλούς συμμετέχοντες. Προσβλέπουμε λοιπόν στην ενεργή συμμετοχή τη δική σας και σε περαιτέρω συζήτηση όσον αφορά την έκθεση αυτή. Πρόεδρος. Πολύ ωραία. Αν υπάρχουν ε, συνάδελφοι που θέλουν να πάρουν το λόγο, στο κάνουν σήμερα το απόγευμα μετά το διάλειμμα, σας παρακαλώ πολύ. Ναι, μπορείτε να μιλήσετε σήμερα το απόγευμα. θα είμαι πολύ σύντομη. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλή η γνωμοδότηση, γιατί από τι περιστάσει ε, στον περιορισμένο χώρο που είχε, ε, νομίζω συμπέραμε πολύ σημαντικά θέματα όσον αφορά την καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων γυναικών σε αναπτυσσόμενε χώρε. Οπωσδήποτε με τις τροπολογίες μας θα αναφέρουμε τις άλλες περιοχές που έχει θίξει η κυρία Σέσκοβα όσον αφορά την ενδυνάμωση των γυναικών, ε, των αλφαβητισμών τους, γιατί υπάρχει και πρόβλημα ε, με αναλφαβητισμό των γυναικών και οπωσδήποτε η άγνοια και η αλλαγή της κουλτούρας, των στερεοτύπων είναι κάτι το οποίο μπορεί να βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τέτοια προγράμματα. Στις δικές μου τροπολογίες θα, συμπεριβα... Ε, θα ενισχύσω αυτά που έχει θίξει ήδη η συγγραφιά της γνωμοδότησης, ε, βάζοντας επιπρόσθετα και άλλες περιοχές όπου μπορούμε να βοηθήσουμε τις γυναίκες να ενδυναμωθούν περισσότερο. Γι' αυτό δεν θα μπορέσω να έρθω το απόγευμα και γι' αυτό ήθελα να πω αυτά τα δύο λόγια. Ευχαριστώ. Tack så mycket för det och jag ber om ursäkt att eh, är så kort tid, men du får ναι. Λυπάμαι πραγματικά που είχαμε τόσο λίγο χρόνο. Έχετε πάλι το λόγο, παρακαλώ. Εισηγήτρια, Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την δυνατότητα που μου δίνετε να συζητήσουμε την γνωμοδότηση αυτή σήμερα το απόγευμα. Σας ζητώ πάντως συγγνώμη γιατί νόμιζα ότι θα συζητούσαμε την γνωμοδότησή μου τώρα το πρωί. Εγώ δεν θα είμαι σε θέση να έρθω το απόγευμα στην Επιτροπή μας. Πρόεδρος. Μάλιστα. Σας ζητώ λοιπόν συγγνώμη. Σας ζητώ συγγνώμη που αφαιρώσαμε τόσο λίγο χρόνο στη γνωμοδότησή σας σήμερα το πρωί. Ειλικρινά, σας ζητώ συγγνώμη λοιπόν. Πρέπει να ολοκληρώσουμε πάντως στο σημείο αυτό τη συζήτησή μας και να διευκρινίσω το εξή. Προθεσμία κατάθεση τροπολογιών. 17 Ιουλίου το μεσημέρι, 12 το μεσημέρι, η Επιτροπή μας θα ψηφίσει στις 3 Σεπτεμβρίου και η Επιτροπή Ανάπτυξη στις 18 Σεπτεμβρίου. Και θα περάσει στη συνέχεια στην Ολομέλεια η έκθεση αυτή. Ολοκληρώνουμε λοιπόν το σημείο αυτό και θα ήθελα να σε υπενθυμίσω ότι έχουμε μια σημαντική ψηφοφορία στις 3 όσον αφορά το νομοθετικό πακέτο για τα θύματα. Κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ στις 3 το απόγευμα στην αίθουσα της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Θα συνεχίσουμε πάντως εδώ με τη συνεδρίασή μας στις 3.30. Ο Πρόεδρος ευχαριστεί τους διερμηνείς. Καλό απόγευμα. Καλό μεσημέρι.